På Καλώς ήρθατε στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Σας καλωσορίζω σε αυτήν την δημόσια κρόαση για την κατάσταση των ανήπαντρων μητέρων. Χαίρομαι ιδιαίτερα που καλωσορίζω τόσους συναδέλφους και συμμετέχοντες ε, και καλωσορίζω βεβαίως ε, τις ε, ειδικού μας οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτών που θα συναντήσουμε. Επίσης, καλωσορίζω τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Παρασκευά δηλαδή, από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης η σημερινή ακρόαση για την κατάσταση των ανήπαντρων μητέρων είναι μέρος της εργασίας ε, της Επιτροπής μας. Εμείς αποφασίσαμε να συντάξουμε μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας που θα είναι πάρα πολύ σημαντική και χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να παρουσιάσω την εισηγητριά μας, την κυρία Ματέρα, η οποία έχει δείξει πάρα πολύ μεγάλη αφοσίωση σε αυτό το θέμα. Το σημερινό μας, η σημερινή μας συζήτηση θα γίνει σε δύο μέρη. Το πρώτο κομμάτι έχει ως θέμα τη νέα κατάσταση, τη νέα μορφή των οικογενειών και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ε, τα νοικοκυριά με μία μητέρα, με μία μητέρα, ναι, και το ότι μπορεί να γίνει για να υποστηριχθούν οι ανήπαντρες μητέρες. Βεβαίως οι κοινωνίες μας αλλάζουν, οπότε αλλάζουν ε, και οι μορφές της οικογένειας. Και αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι να εξετάσουμε τις αλλαγές οι οποίες εμφανίζονται στην κοινωνία και να λάβουμε βεβαίως υπόψη ε, τις καλύτερες λύσεις και τις βέλτιστες πρακτικές. Ναι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση στην κοινωνία. Να λάβουμε υπόψη τις νέες καταστάσεις που επικρατούν. Θα ήθελα να πω εισαγωγικά πως ε, γεγονό είναι πως ε, βλέπουμε πάρα πολλές ε, ανήπατρες μητέρες στη σημερινή κοινωνία αλλά πρέπει να θυμόμαστε πως πάντα είχαμε ανήπατρες μητέρες εγώ η ίδια μεγάλωσα με πέντε αδέρφια και μία ανήπαντρη μητέρα που μας ανέθρεψε. Για τον το λόγο ότι η μητέρα μου πέθανε, ο πατέρας μου συγχωρείτε, πέθανε όταν ήμασταν παιδιά. Οπότε έχω προσωπική εμπειρία και ξέρω τι σημαίνει μια μητέρα μόνη. Η μητέρα μου κατάφερε να αναθρέψει έξι παιδιά για να γίνουμε οι πολίτες που είμαστε σήμερα. Και αυτό συμβαίνει... Αυτό συνέβαινε πάντα για διάφορους λόγους. Ο ένας γονιός ε, είχε το καθήκον να αναθρέψει την οικογένεια μόνος του ή μόνη της. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως πως ε, υπάρχει... Αυτό είναι ένα πρόβλημα που χρειάζεται λύση. Δεν είναι πρόβλημα είναι μια συνήθις κατάσταση, έχουμε δει παραδείγματα για το πώς είναι δυνατόν να γίνει, να βγούμε επιτυχώς από μια τέτοια κατάσταση, αλλά του τουλεχθέντος βεβαίως πρέπει η κοινωνία να βοηθάει. Αυτά λοιπόν εν είδη εισαγωγής ε, για ένα πολύ ενδιαφέρον ελπίζω απόγευμα, το οποίο θα αυξήσει τις γνώσεις μας και ελπίζω όλοι μαζί να μπορέσουμε να, εξετάσουμε και να βρούμε λύσεις στην κατάσταση που αντιμετωπίζουν αυτές οι οικογένειες. Οπότε σας καλωσορίζω και πάλι θερμότατα και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα δώσω τον λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Ματέρα. θα κάνει μια εισαγωγή. Έχετε λοιπόν το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ, όπως η Πρόεδρος, να χαιρετήσω τους προσκεκλημένους μας, τους εξαιρετικούς εμπειρογνώμονες και τους πολυάριθμους και πολυάριθμους συναδέλφους που βρίσκονται σήμερα στην αίθουσα. Σήμερα θα αρχίσουμε να εξετάζουμε ένα θέμα, το θέμα των ανήπαντρων μητέρων, ένα θέμα που είναι αρκετά παλιό. Αλλά σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε να το συζητήσουμε. Και οφείλουμε να το συζητήσουμε και αυτή η συνάντηση σήμερα με την παρουσία των εμπειρογνωμόνων είναι η καταλληλότερη ευκαιρία για να βρούμε συγκεκριμένε λύσει και στο το δυνατόν συντομότερα. Η Επιτροπή των Δικαιωμάτων των Γυναικών και τη Ισότητα των Φίλων στο Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει συγκεκριμένα να αρχίσει να ασχολείται με το πρόβλημα, με το ζήτημα αυτό. Πρέπει να πω ότι τα στατιστικά δεδομένα προκαλούν ε, ανησυχία τους τελευταίους μήνες, γιατί ο αριθμός των ανήπαντρων ιτέρων ε, τις τελευταίες, ε, τους τελευταίους μήνες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας αυξάνεται διαρκώς. Και αυτό είναι μια πραγματική αναπηρία, η ένδυα. Οι γυναίκες αυτές όχι μόνο είναι ανήπαντρες και μόνες, αλλά και φτωχές, κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτό γίνεται ένα ακόμη λόγο για διακριτική μεταχείριση. Οι γυναίκε είναι πιο φτωχέ από ότι οι άντρε. Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα των στατιστικών ε, μελετών που μα τα επιβεβαιώνει και η έκθεση για την κατάσταση των μητέρων και των ε, παιδιών, την ε, έκθεση που λάβαμε πρόσφατα και που αποδεικνύει πόσο ο αριθμός των γυναικών αυτών, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο αυξάνεται και μάλιστα δραματικά. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει λοιπόν εδώ να τοποθετηθεί. Να τοποθετηθεί με σαφήνεια και αποφασιστικότητα όσο το δυνατόν συντομότερα. Γι' αυτό η πρόεδρος Σπέντσον σωστά υπογράμμισε ότι βρισκόμαστε εδώ για να συλλέξουμε τις παρατηρήσεις των εμπειρογνωμόνων και να ακούσουμε τις απόψει τους, για να αρχίσουμε να ξεφυλίζουμε τις σελίδε αυτή τη έκθεση τις οποίες αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή να είμαι εισηγήτρια. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, διότι ως Ιταλίδα θα μπορούσα να φλιαρίσω. Αλλά εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο έμαθα να εκφράζομαι κάπως πιο σύντομα, με ακρίβεια και πιο συνοπτικά, ώστε να φτάνω κατευθείαν στον πυρήνα των ζητημάτων για να είμαστε όσο δυνατόν πιο αποτελεσματικέ και ε, να φτάνουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Εμείς οι γυναίκες ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να είμαστε συγκεκριμένες και αποτελεσματικές. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να δώσω αμέσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες του πρώτου πάνελ. Ο τίτλος του πρώτου πάνελ, τη πρώτη ομάδα συζήτηση που θα συζητήσουμε και θα εξετάσουμε εντελεχώ, είναι το νέο πρότυπο τη οικογένεια και οι προκλήσει που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ανήπαντρε γυναίκε. Οι δύο εμπειρογνώμονε είναι η καθηγήτρια Ρωσάνα Τριφιλέτη, καθηγήτρια κοινωνιολογίας και θεμάτων οικογένεια και κοινωνικών πολιτικών στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας στην Ιταλία και η δόκτωρα Λιπράντη, η οποία είναι διευθύντρια ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο για, την, για τις Κοινωνικές Έρευνες στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Ξεκινάμε κατευθείαν λοιπόν με την κυρία Τρίφιλέτη, καθηγήτρια κοινωνιολογίας για θέματα οικογένειας και κοινωνικών πολιτικών. Έχει πολλές δημοσίευσεις στο ενεργητικό της για τα θέματα αυτά, ιδίως για όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κατάσταση των ανήπαντρων μητέρων. Ήθελα απλώς να πω στην εμπειρογνώμονά μας ότι έχουμε 15 λεπτά στη διάθεσή μας μόνο. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Δεν θα μιλήσω στα αγγλικά γιατί εκφράζομαι καλύτερα στη μητρική μου γλώσσα. Ε, ε, ε, θα προσπαθήσω το να παρουσιάσω τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις ανήπαντρες μητέρες. Ως ανήπαντρη μητέρα και εγώ ίδια αισθάνομαι ότι τα ζητήματα αυτά με αφορούν ιδιαίτερα. Έχω ζήσει την εμπειρία του διαζυγίου και του μετέπειτα μοναχικού βίου. Αλλά καθότι είμαι ακαδημαϊκός θα ξεκινήσω πρώτα από το ζήτημα θεωρητικά και από τα όρια των γνωσεών μας για το συγκεκριμένο θέμα. Θα ήθελα να δώσω έμφαση στο εξής. Δεν πρέπει καθόλου να έχουμε τυφλή εμπιστοσύνη στα στατιστικά δεδομένα. Γιατί αυτό που συχνά περιγράφουν τα στατιστικά δεδομένα στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο αξιόπιστο όσο τα αποτελέσματα των ποιοτικών ερευνών που γίνονται στην πράξη, επιτόπου. Ε, ως κοινωνιολόγος Πρέπει να πω ότι εδώ και 15 χρόνια κάνω έρευνες για το θέμα αυτό, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της ποιοτική κοινωνιολογίας. Και βρίσκονται τα αποτελέσματα αυτού του είδους των ερευνών, του δεύτερου, τελικά είναι και πιο πιστικά και περισσότερο αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα σε σχέση με τα αφηρημένα δεδομένα των στατιστικών, που πολύ συχνά πρέπει να τα αναλύει κανείς μόνο εντός ενός συγκεκριμένου πλαισίου. Ως ανήπαντρη μητέρα, καμία γυναίκα δεν ε, είναι τελείως ε, απελευθερωμένη και από τις στατιστικές παραδόσεις της κάθε χώρας. Το φαινόμενο, όπως είπαν και οι προλαλήσασες, είναι γενικευμένο, αλλά δεν σημαίνει ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χωρών. Θα προσπαθήσω λοιπόν να διορθώσω την παρουσίασή μου γύρω από τα βασικά αυτά σημεία. Και θα προσπαθήσω να αναπτύξω αυτές τις πτυχές, προσπαθώντας ταυτόχρονα να κάνω κάποια σχόλια και για τον προβληματισμό που έχει να κάνει με την αιτιολογία της ε, κατάστασης του μοναχικού γονέα, του γονέα που είναι ανήπαντρος ή και της φτώχειας. Η φτώχεια βεβαίως κάνει πιο ευάλωτο, πιο ε, εκτεθειμένο τον, μοναχικό, το μόνο γονέα από ότι αυτόν που ανήκει σε μια οικογένεια. Μιλάμε για τις οικονομικές συνθήκες εδώ. Θα προσπαθήσω μάλιστα να ολοκληρώσω καταλήγοντας να εντοπίσω, επειδή είχα την τύχη να ετοιμάσω για την Επιτροπή DG5 ε, ε, απασχόλησε κοινωνικά προβλήματα, μια έρευνα, μια μελέτη το 2007, που ήταν μια συγκριτική μελέτη για 13 χώρες. Η έκθεση αυτή ασχολείται με το θέμα της φτώχειας αυτού του είδους της οικογένειας. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορούσα να αποτολμήσω και να δώσω κάποιες ιδέες για το πώς μεταβάλλονται οι πολιτικές των ευρωπαϊκών κρατών σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα και θα επιχειρήσω να διατυπώσω και κάποιες συστάσεις για το ποια κατεύθυνση θα ήταν καλό να ακολουθήσουν οι πολιτικές μας προτάσεις. Και αυτό γιατί είναι και πολύ δύσκολο να εξηγήσει κανείς τα αίτια του φαινομένου αυτού βάσει μια συγκεκριμένη οικογενειακή δομή και μόνον. Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε συνέστηση ότι ακόμη και τα δεδομένα Eurostat έχουν μια σχετική σύγκληση, αλλά δεν περιγράφουν πάντοτε ακριβώς το ίδιο φαινόμενο όταν μιλούμε για μόνους γονείς, μονογονεϊκές οικογένειες. Αυτό εξαρτάται και από την ε, πολιτιστική παράδοση της κάθε χώρας. Ο, υπάρχουν χώρες όπου το κλασικό οικογενειακό μοντέλο είναι τόσο ισχυρό σε πολιτιστικό επίπεδο, στο επίπεδο της νοοτροπίας, που τίνει κανείς να ορίζει την μονογονεϊκή οικογένεια ως μια απόκληση σε σχέση με τον γενικό κανόνα. Ξεχνάνε δηλαδή πολλές φορές ότι υπάρχουν πολλές μορφές οικογενειών και ότι υπάρχουν διαφορές σε πολιτιστικό επίπεδο κατά κύριο λόγο. Αυτό γίνεται φανερό με πολλές διαφορετικές εκφάνσεις. Να δώσω ένα απλό παράδειγμα. Πρόσφατα στον Ολλανδικό τύπο διάφασα πάλι ένα άρθρο όπου λέγεται ότι οι γυναίκες δεν θα πρέπει να υποχρεώνονται για οικονομικούς λόγους να μην ε, μπορούν να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους την ε, συνδρομή μια τροφού. Αυτά θα προσπαθήσω να αναλύσω. Πρώτα απ' όλα τι ε, εννοούμε με τους ανήπαντρους γονείς σε διάφορες χώρες. Αυτό εξαρτάται πάντοτε από τα διαζύγια και τα ποσοστά γεννήσεων εκτός γάμου. Αυτά έχουν αυξηθεί βεβαίω σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά με ρυθμούς αύξηση διαφορετικούς. Στην Ευρώπη τη δεκαετία του 2000 τριπλασιάστηκαν οι γεννήσεις εκτός γάμου, αλλά στη Γαλλία τετραπλασιάστηκαν, ενώ τριπλασιάστηκαν στην Ιταλία, στην ε, Σουηδία που όλοι θεωρούμε πιο προχωρημένοι σε αυτά τα ζητήματα, εκεί η αύξηση είχε γίνει σε προηγούμενα χρόνια. Θα πρέπει κανείς επίσης να φανταστεί ότι θα πρέπει να είμαστε σε θέση να διακρίνουμε οικογένειες μονογονέικες, de jure de facto, βάσει του νόμου δηλαδή, λόγω των πραγματικών συνθήκων. Εάν δούμε πώς λειτουργεί μια οικογένεια από αυτήν την προοπτική, από αυτή την οπτική γωνία και όχι μόνο τους επίσημους θεσμούς του γάμου και των ε, ζευγών που συμβιώνουν θα αντιληφθούμε ότι υπάρχουν ίσως ακόμη περισσότερες μορφές οικογενειών ε, μονογονεϊκών και σε σχέση με τα ζευγάρια στην καθημερινή τους λειτουργία. Γιατί κάποιες επισήμως μονογονεϊκές οικογένειες καταλήγουν ε, σε οικογένειες που απλά συμβιώνουν. Αυτό εξαρτάται από την ομοθεσία διαβόρων χωρών και το αν ε, κυρώνουν επισήμου το καθεστώ μια ε, οικογένεια που το ζεύγο των γονέων απλώ συμβιώνει. Ο προβληματισμός προβληματισμό αυτών των μεθόδων και των τρόπων να καταμετρά κανεί το φαινόμενο οδηγεί στα εξή. Βλέπει κανεί όρια ηλικιακά διαφορετικά από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν χώρε όπω η Ιταλία που θεωρούν μονογονική οικογένεια την οποιαδήποτε οικογένεια χωρί κανένα ηλικιακό όριο. Δηλαδή ένας ε, κύριος 80 χρονών που έχει ένα γιο 60 θεωρείται μονογονεϊκή οικογένεια. Άλλες χώρες έχουν όρια όπως τα 16, τα 18, τα 25, τα 26. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ιδιαίτερα αξισημείωτη διαφορά στην καταμέτρηση. Πραγματικά έχουν γίνει προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο να παρακολουθηθεί αυτή η ποικιλία, οι τόσες διαφορές, αλλά βρισκόμαστε στα πρώτα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Πάνελ και πηγαίνουμε λίγα χρόνια πίσω σε αυτά τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Πάνελ. Με τα χρόνια που έχουν περάσει δεν έχουμε ακόμη αξιόπιστα αποτελέσματα σύγχρονα, επικαιροποιημένα τα οποία να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως σημείο αναφοράς. Σε αυτές τις διαφορές της καταμέτρησης πρέπει να σκεφτούμε ότι έρχονται να προσθεθούν και διαφορές δημογραφικές. Δηλαδή, μέσα σε μια χώρα μπορεί να υπάρχει ένα πιο έντονο φαινόμενο προορισμητρότητας, δηλαδή των εφήβων που γίνονται μητέρες. Στην ε, Αγγλία κυρίως, στις αγγλώσσακισμικές χώρες και μάλιστα στην Ουαλία, η πρόορη μητρότητα και οι έφηβες μητέρες είναι ένα γεγονός που επηρεάζει ιδιαίτερως και το φαινόμενο της μονογονεϊκής οικογένειας. Μιλάμε για οικογένειες με συγκεκριμένα προβλήματα, με πολύ νέα παιδιά και βεβαίως αυτό πολλές φορές συνδυάζεται με ένα υψηλό ποσοστό διαζυγίων. Και τα παιδιά θα πρέπει να υποστούν τις ε, συνέπειες αυτές σε μεγαλύτερη ηλικία. Εδώ το θέμα δεν είναι απλώς η αριθμητική αύξηση αυτού του είδους των οικογενειών που υποδεικνύει ότι υπάρχει ένα θέμα με την όλη κατάσταση. Αυτό που ενδιαφέρει είναι τι δυνατότητες προσφέρουν οι κοινωνικές πολιτικές αυτές τις οικογένειες. Αυτό δίνει πολλέ διαφορές και έτσι καταλήγουμε σε ποσοστά φτώχεια πολύ διαφορετικά ανάλογα με τα είδη οικογενειών ε, μονογονεϊκών. Έτσι υπάρχουν χώρες όπου έχουμε ψηλότατα ποσοστά σε σχέση με τις κλασικές οικογένειες για τις μονογονεϊκές όπως η Σουηδία και η Νορβηγία, αλλά εκεί έχουμε χαμηλά ποσοστά φτώχεια για τι συγκεκριμένε αυτέ τι οικογένειε, διότι η κρατική παρουσία μειώνει τον κίνδυνο φτώχεια. Εάν συγκρίνουμε την οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης ως προς τις κανονικές και τις μονογονεϊκές οικογένειες, αλήθεια είναι ότι καταλήγουμε σε κάποια φαινόμενα που επαναλαμβάνονται. Ιδίω ό,τι αφορά την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Διότι οι οικογένειες, οι μονογονεϊκές, από άποψη αριθμητική, είναι ως επιτοπλίστων φτωχότερες από τις οικογένειες που έχουν ένα ζεύγος γονέων. Κάποια παραδείγματα από τη Eurostat που πρέπει να, βέβαια να τη βλέπουμε επιφυλακτικότητα για όλους τους λόγους που είπα πριν. Οι συνθήκες διαβίωσης των μογονεικών οικογένειών έχει μειωθεί κατά 11% και 23% σε σχέση με οικογένειες με έναν γονιό που εργάζεται και 27% σε σχέση με οικογένειες που έχουν δύο γονείς που εργάζονται. Αυτά προφανώς καταλήγουν, δίνουν πολύ διαφορετικά αποτελέσματα για τις ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ τους. Έτσι, ξέρουμε ότι στη Γαλλία ένα στα τρία παιδιά που ζουν σε μονογονεϊκή οικογένεια, κάτω από το όρο της φτώχειας, μάλλον απειλούνται από την φτώχεια ή βρίσκονται κάτω από το όρο της φτώχειας, ενώ στην Αγγλία το η αναλογία είναι παιδιών προς φτώχεια Αν δούμε λοιπόν το όλο πρόβλημα αυτό από την οπτική γωνία των παιδιών, τη φτώχεια των παιδιών, τότε το πρόβλημα οξύνεται ακόμη περισσότερο. Είναι πολύ ευρύ Είναι διαφορετικά αν κάνουμε τις μετρήσεις μας στα παιδιά από ό,τι στους ενηλίκους. Και τώρα για την ε, μελέτη που υπενήχθηκα προηγουμένως με τις 13 ευρωπαϊκές χώρες, εκεί μετρήθηκε για πρώτη φορά ότι δεν είναι και τόσο σίγουρο ότι οι μονογονεϊκές οικογένειες όπου ο μόνος γονέας είναι πατέρας δεν είναι και τόσο φτωχές όσο πιστεύαμε πριν από λίγα χρόνια. Στην πραγματικότητα Είναι πολύ πιο σπάνιο βέβαια να υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες με έναν γονέα που είναι ο πατέρας. Αλλά σε μερικές χώρες όπως τις σκανδιναβικές αυτό αρχίζει να συμβαίνει όλο και περισσότερο. Τελικά λοιπόν καταλήγουν και οι πατεράδες αυτών των οικογενειών να είναι τόσο φτωχοί όσο οι υπόλοιπες μονογονεϊκές οικογένειες. Για γονείς λοιπόν Μόνος. Εδώ είναι πολλά τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν. Ε, η φτώχεια, ο αποκλεισμό, η απομάκρυνση από την αγορά εργασία, ένα φαύλο κύκλος. Έλλειψη πρόσβαση στην εκπαίδευση, αυτό ιδιαίτερο στην περίπτωση των ε, ανήπαντρων μητέρων, που είναι και νέες. Υπάρχει λοιπόν μια ροπή προς την γενικότερη επιδείνωση της κατάστασής τους. Σε σχέση με αυτήν την κατάσταση που προσπάθησα λοιπόν να απεικονίσω και που μας δίνουν τα στατιστικά δεδομένα, τι μπορώ να πούθηκα εγώ από τόσα χρόνια έρευνας με λεπτομερείς συνεντεύξεις, με μητέρες νέες και μόνες που με βοήθησαν πολύ. Το πρώτο βασικό συμπέρασμα είναι ότι πολλές φορές το πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε μετά την ε, λήξη του όλου θέματος. Δηλαδή, εντοπίζουμε το πρόβλημα στις γυναίκες αυτές αφού έχουν υποστεί την προσωπική τους εμπειρία και τις συνέπειες της κοινωνικής πολιτικής της κάθε χώρα Σε όλες τις χώρες όπου υπάρχει ευαισθησία για τα προβλήματα των μονογονεϊκών οικογενειών Και το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλε τι χώρε, στη δική μου λόγω χάρη και τι άλλε μεσογειακέ. Εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει τάση να προσφέρεται κοινωνική συνδρομή Οπότε αυτό επηρεάζει και την κατάσταση των μονογονεϊκών οικογενειών. Τώρα, αν δούμε τα πράγματα από τη γεωγραφική τους άποψη, βλέπουμε ότι πολύ συχνά ξεχνάμε ότι η κατάσταση των μονογονεϊκών ε, οικογενειών, τον ένα είναι κανείς δηλαδή μόνος γονέας, είναι απλώς μια φάση στο βίο του ανθρώπου. Μια περίοδος χρονική. Δεν είναι μια ετικέτα, μια κοινωνική ετικέτα όπως ήταν στο παρελθόν ούτε και αυτό που μας θύμισε πριν ε, η πρόεδρος. Αυτό ισχύει όλο και περισσότερο για τις γυναίκες, για τον βίο των γυναικών, αλλά αρχίζει να ισχύει και για τον βίο των ανδρών. Ένα άλλο πλεονέκτημα από την χρήση των ποιοτικών δεδομένων είναι ότι κατευθείαν βλέπουμε να περιγράφεται η κατάσταση και ενδεχόμενες αποκρίσεις που βρίσκουν οι οικογένειες αυτές τα προβλήματά τους, κάτι που εν μέρη γίνεται χάρη στις κοινωνικές πολιτικές, αλλά και με την ανεπίσημη συνδρομή και στήριξη. Οι φτωχότερε οικογένειε σε διάφορε χώρε μάλιστα, ε, επειδή δεν έχουν ακριβώ πρόσβαση στι κοινωνικέ πολιτικέ, γιατί ακριβώς βρίσκονται σε συνθήκες ανεργίας, επειδή δεν μπορούν να έχουν φρεολογικές ελαφρύνσεις, μα οδηγούν να θέσουμε το εξή πρόβλημα. Μια κοινωνική πολιτική που πρέπει να λάβει υπόψη σε όλο αυτόν τον προβληματισμό δεν θα πρέπει να λάβει υπόψη και την διατήρηση αυτών των αυθόρμητων δικτύων κοινωνικών ομάδων που δημιουργούνται γύρω από τι οικογένειε που έχουν ε, ανάγκη. Ε, αυτό ισχύει πάρα πολύ για το μεσογειακό σκηνικό και τοπίο. Στην Ισπανία, την Πορτογαλία, πολλές φορές Μοιάζει να υπάρχουν λιγότερε οικογένειε μονογονεϊκέ, γιατί αμελού, παραμελούμε το γεγονό ότι οι οικογένειε με έναν γονέα στη Μεσόγειο αποτελούν μέρο μια ευρύτερη οικογένεια. Ζουν στα πλαίσια μια διευρυμένη οικογένεια. Απλώ δεν τι εντοπίζουμε λοιπόν. Αυτού του είδου η συνδρομή, η βοήθεια θα μπορούσε. Θα μπορούσε λοιπόν να προβληθεί περισσότερο και να υποστηριχθεί. Ένα άλλο πλεονέκτημα από την χρήση των ποιοτικών μελετών είναι ότι μπορούμε να δούμε τον άμεσο αντίκτυπο των πολιτικών και μπορούμε έτσι να προβάλλουμε και μελλοντικέ πολιτικές και να τις σχεδιάσουμε βασιζόμενοι στις αυθόρμητες τάσεις που υπάρχουν στα πλαίσια αυτών των οικογενειών. Όπως η μεγάλη αυτή επιθυμία να έχει κανείς πρόσβαση στην επίσημη αγορά εργασίας. Αυτό ίσως είναι το ζωτικότερο σημασία θέμα για τις οικογένειες αυτές. Θα μπορούσε κανείς επίσης να σχεδιάσει πολιτικές που αντιμετωπίζουν και καλύπτουν τις ανάγκες αυτού του είδους των οικογενειών. Κάτι άλλο που βλέπουμε ξεκάθαρα είναι ότι ένα μεγάλο μέρος, ιδίω στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, ένα μεγάλο μέρος των πολιτών, βλέπουν οικογένειε που δεν βρίσκονται στην επίσημη αγορά εργασία να δουλεύουν παρόλα αυτά στη μαύρη αγορά. Ιταλία και η Ελλάδα έχουν ένα μεγάλο μέρος από 25-30% του ΑΕΠ που παράγεται ακριβώς από αυτή την παραοικονομία. Άρα και αυτό είναι ένα πολύ σαφές δεδομένο και κάτι άλλο που προκύπτει με σαφήνεια από τις ποιοτικές μελέτες είναι ότι ένας γονέας που μόνος μεγαλώνει τα παιδιά του συμπυκνώνει στο πρόσωπό του τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κανείς το να συνδυάσει τον επαγγελματικό βίο με την ε, ανατροφή των παιδιών. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κατεπηγόντως διότι συνδέει αυτό τις μονογονεϊκές οικογένειες με τον γονέα να εργάζεται μόνο στη μαύρη αγορά ή σε παράνομες, παράτυπες μορφές εργασίας. Ε, εκεί βλέπουμε να συνδυάζεται αυτό με, το, με την απώλεια του κοινωνικού μας κεφαλαίου, ενός ε, μεγάλου ε, κεφαλαίου γνώσης και εμπειρίας και εκπαίδευσης. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να εξοικονομήσουμε ό,τι μπορούμε. Ήθελα να παρουσιάσω απλώ ορισμένα ζητήματα για τα οποία ακόμη δεν γνωρίζουμε αρκετά. Είναι απαραίτητο να κάνουμε καθεαυτή κοινωνιολογική έρευνα διότι η Ευρώπη θα μπορούσε να οργανώσει μια τόσο δαπανηρή έρευνα. Όχι μόνο δείγματα πλέον, όχι μόνο δειγματοληπτικά, αλλά σε όλες τις χώρες και τις 27 και ακόμη και σε αυτές που έχουν κάνει αίτηση για την προσχώρησή του. Για την ένταξή του, Η έρευνα αυτή θα έπρεπε να επικεντρώνεται ενδεχομένω στο στο ποιε πολιτικέ, γιατί λειτουργούν καλύτερα και γιατί στα δεδομένα, στις δεδομένες συνθήκες λειτουργούν καλύτερα. και πώς επιτρέπουν να γίνεται η μετάβαση ή ο συνδυασμός μεταξύ των, ε, της φροντίδας των παιδιών, της ανατροφής των παιδιών που κάποιος μπορεί να τα παρακολουθεί και του επαγγελματικού βίου, αυτό, αυτό ιδίως για τις γυναίκες. Καταλήγω κάπως σύντομα στο συμπέρασμά μου σε σχέση με τα αποτελέσματα των χωρών που ανέφερα προηγουμένως. Εγώ νομίζω ότι ήδη έχει ξεκινήσει μια διαδικασία όπου υπάρχει μια σχετική σύγκληση των κοινωνικών πολιτικών στην Ευρώπη, οπότε χώρες που προηγουμένως και με πιο με περισσότερη ανάγκη έπρεπε να αντιμετωπίσουν, περισσότεροι έπρεπε να αντιμετωπίσουν το θέμα των γονεϊκών οικογενειών, τώρα έχουν αρχίσει να ξανασχεδιάζουν την κοινωνική τους πρόνοια προς την σωστή κατεύθυνση. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα και που είναι έμπλεο συμβολικών μηνυμάτων είναι το να βάλουμε σε χρονολογικό κατάλογο τις χώρες που έχουν ξεκινήσει αυτή την μεταρρύθμιση των πολιτικών τους. Αλλά το ίδιο θα μπορούσαμε να κάνουμε και με τις χώρες που άρχισαν να μεταβάλουν την κοινωνική τους προστασία ως από προστασία που έκανε διάκριση έκανε διάκριση στην πολιτική της ως προς τους γονείς και έχει εγκαταλείψει τα επιδόματα χειρίας ορφανών αλλά κατευθύνεται πλέον σε μια γενίκευση της αντιμετώπισης του φαινομένου των μονογονεϊκών οικογενειών. Γιατί μόνος γονές μπορεί να είναι κανείς λόγω χειρίας, λόγω διασγείου. Οι συστάσεις μου, σε αυτές να επιστρέψω μετά, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, θα ήταν ακριβώς αυτές. Δηλαδή, μια από τις μετρήσεις που θα έπρεπε να κάνουμε και που πρέπει να προαγγείλω και να παροτρύνω να γίνει, είναι χώρες που δεν έχουν ακόμα αυτή την πρόβλεψη ε, για τις μονογονεϊκές οικογένειες να προσφέρουν ένα επίδομα στην περίπτωση που ο πατέρας στο μεταβόδιαζίκιο δεν μπορεί να προσφέρει διατροφή. Ευχαριστούμε την καθηγήτρια Τριφυλέτη για όσα μας είπε. Να δώσουμε αμέσω το λόγο στην δεύτερη εμπειρογνωμονά μας αυτής της ομάδας προσκεκλημένων την κυρία Λάουρα Αλιπράντη, διευθύντρια ερευνήτρια του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Είναι μέλος της ΚΕΤΗ, της Επιστημονικής Επιτροπής για Έρευνα Θεμάτων σε σχέση με την Ισότητα των Φύλων και έχει ασχοληθεί με το συντονισμό πολλών ερευνητικών μελετών σε σχέση με την ισότητα των φίλων, τις κοινωνικές πολιτικές και τις οικογένειες. Θα ζητούσα από την δόκτωρα να ε, παραμείνει λίγο στο όριο του χρόνου ομιλίας γιατί έπειτα δεν θα μπορέσουν να παρέμβουν οι συνάδελφοι. Θα θέλαμε λοιπόν λίγο χρόνο και για την ίδια τη συζήτηση. Ευχαριστώ. thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο καθώς επίσης και τα μέλη της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Φίλων που με προσκάλεσαν σε αυτή τη δημόσια ακρόαση. Είμαι η δεύτερη σε σειρά ομιλήτρια. Θεωρώ λοιπόν ότι κάποια πράγματα ήδη έχουν υποθεί από την κυρία Ροζάνα Τριφιλέτη, η οποία πήρε πρώτα το, πήρε πρώτη το λόγο. Ε, συγχωρήστε με λοιπόν αν επαναλάβω κάποια πράγματα. Από τη δεκαετία του 60 και μετά έχουν γίνει πολλές αλλαγές. Πολλές αλλαγές στο μοντέλο της δημιουργίας της οικογένειας, της απόκτησης των παιδιών, καθώς επίσης και της διάλυσης οικογένειας. Έχουμε ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό γάμων, μία αύξηση στο, στην ηλικία κατά την οποία παντρεύεται κανείς ή που αποκτά παιδιά. Επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει μία μείωση στην, στο μέσο μέγεθος της οικογένειας καθώς επίσης και μία αύξηση στις γεννήσεις εκτός γάμου. Επίσης έχουμε νέες μορφές οικογένειας, ένωση με συγκατάθεση συμβίωση, νοικοκυριά ενός ατόμου, μονογονεϊκές οικογένειες, επανασυσταθήσεις οικογένειες κτλ. Επίσης ο έγαμος βίος έχει γίνει πιο εύθραστος και φαίνεται ότι οι κοινωνικές δομές και τα πρότυπα έχουν αντισταθεί στον πλουραλισμό των επιλογών που υπάρχουν πλέον στην διαμόρφωση ζευγαριών. Στην Ευρώπη έχουμε όλο και περισσότερα ζευγάρια τα οποία ζουν σε καθεστώς συμβίωσης και πάρα πολλοί γάμοι καταλήγουν πλέον σε διαζύγια. Επομένω, ο γάμο και η ιδιότητα του γονέα όλο και περισσότερο είναι έννοιε οι οποίε δεν συνδέονται μεταξύ του. Βλέπουμε ότι η συγκατοίκηση πολλές φορές είχε καταστήσει τον γάμο και πολλά ζευγάρια δεν είναι επαντρεμένουν να αποκτούν το πρώτο τους παιδί. Μια σημαντική αλλαγή είναι ένα σημαντικό φαινόμενο είναι η αύξηση των γεννήσεων εκτός γάμου. Πιο συγκεκριμένα, το 2009 περίπου 35% όλων των παιδιών στην Ευρώπη γεννήθηκαν ε, έξω από τα επίσημα δεσμά του γάμου. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει το ποσοστό αυτό. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Επίσης υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις διάφορες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως υπόθηκε άλλωστε στις σκανδιναβικές και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες έχουμε τα υψηλότερα ποσοστά. Περίπου 50% των παιδιών γεννιούνται εκτός του επίσημου γάμου, ενώ στην κεντρική Ευρώπη το ποσοστό αυτό είναι γύρω στο 40%. Το νέο όμως φαινόμενο που έχουμε είναι ότι ε, στις νότιες ευρωπαϊκές χώρες έχουμε μια σημαντική αύξηση στο ποσοστό αυτό. Ωστόσο, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα, για παράδειγμα, το ποσοστό είναι αρκετά χαμηλό, πολύ χαμηλό, 7% μόνο. Βέβαια υπάρχουν κάποιες κοινωνικές προκαταλήψεις για την ανήπαντρη μητέρα, καθώς επίσης και απουσία οποιασδήποτε πολιτικής υποστήριξης από το κράτος και αυτά με τη σειρά τους συμβάλλουν στον μικρό αριθμό γάμων εκτός γάμου. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και αυτό το μικρό ποσοστό στην Ελλάδα, 7% όπως σας είπα. Υπάρχουν κάποια προβλήματα με τους ορισμούς όμως τώρα. Όσον αφορά τις μονογονεϊκές οικογένειες, η καθηγήτρια Τριφυλέτη αναφέρθηκε σε αυτά. Υπάρχουν ε, κάποιες δυσκολίες μέτρησης όσον αφορά τα ποσοστά μονογονεϊκών οικογενειών. Ποιο νοικοκυριό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μονογονεϊκή οικογένεια. Υπάρχει πάντα το θέμα των εξαρτώμενων παιδιών, της εξάρτησης, της συντήρησης των παιδιών από τον γονέα. Επομένως, η μονογονεϊκή οικογένεια είναι η οικογένεια που έχουμε έναν ενήλικο γονέα και τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο ενήλικο παιδί. Βέβαια το ζήτημα της εξάρτησης αυτής της συζήτησης, ε, της συντήρησης με συγχωρείτε, αποτελεί αντικείμενο περισσότερης ανάλυσης όσον αφορά τον κατάλληλο ορισμό. Η Eurostat ε, αντιμετωπίζει τα εξαρτώμενα παιδιά με βάση κάποιες ηλιακές ομάδες, 16 έτη, 16 με 24 έτη ή τουλάχιστον τα παιδιά εκείνα τα οποία ζουν σε οικογένειες με έναν γονέα, ο οποίος θεωρείται ότι είναι οικονομικά μη ενεργός. Κάτι το οποίο αναφέρθηκε και πριν από λίγο είναι η περίπτωση των μόνων γονέων με ένα παιδί ανήλικο που συνεχίζουν και ζουν οι ίδιοι με τους γονείς τους. Το μοντέλο αυτό το βλέπουμε συχνά σε χώρες της Νότιας Ευρώπης. Περίπου το 2% των, του συνόλου των νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβάνουν και μία μόνο οικογένεια. Σύμφωνα με κάποια πρόσφατα στοιχεία βλέπουμε ότι ε, τα μόνο γωνιακά νοικοκυριά αντιστοιχούν περίπου στο 13% του συνόλου των ιδιωτικών νοικοκυριών με παιδιά στην Ευρώπη των 25-2005. Αντίστοιχα ποσοστά είναι για το Βέλγιο 18%, Εστονία 17%, Δανία και Γερμανία 16%, 5% μόνο στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα, όπου βλέπουμε, όπως βλέπετε, τα χαμηλότερα ποσοστά. Οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι το 90% των μόνων γονέων και πάλι εδώ πέρα υπάρχουν διαφορές από τη μια χώρα στην άλλη. Τα υψηλότερα, υψηλότερα ποσοστά είναι στην Ιρλανδία, ακολουθεί η Αυστρία, η Γερμανία στην Ελλάδα είναι 91% το αντίστοιχο ποσοστό. Οι περισσότερες μόνες μητέρες ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 30 με 39 ε, έτη. Βλέπετε εδώ πέρα πάλι τις διαφορές ανάμεσα στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε πιο νέες μόνες γυναίκες μητέρες στον Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Μάλτα. Εκείνοι οι χώρες λοιπόν όπου οι μόνες μητέρες είναι νεότερες. Έχουμε τρεις ε, κατηγορίες μόνον ε, γυναικών, μόνες γυναίκες αδίπαντρες ή εξαιτία χειρίας ή, ή λόγω διαζυγίου. Βλέπετε εδώ πέρα ότι ε, έχουμε διαφορετικές καταστάσεις και επομένως χρειαζόμαστε και διαφορετικές πολιτικές και διαφορετικά μέτρα υποστήριξης. Θεωρούμε ότι το πιο συχνό φαινόμενο είναι αυτό των μόνων γυναικών εξαιτία διαζυγίου. Βλέπουμε όμως πάλι ότι σε πάρα πολλές χώρες τα ποσοστά των ε, διαζευμένων γυναικών ε, είναι τα ίδια με τα ποσοστά των ε, ανήπαντρων γυναικών. Τα νοικοκυριά με μόνες μητέρες είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε διάφορα κοινωνικά φαινόμενα και επίσης δεν έχουν την απαραίτητη κοινωνική υποστήριξη, γιατί καλούν αστικά να καλύψουν δύο ρόλους, εργασία και φροντίδα για τα παιδιά. Η βασική επίπτωση εδώ πέρα εξαρτάται από την πραγματική συμβολή του πρώην συντρόφου, της, του πατέρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς επίσης και από την υποστήριξη που υπάρχει από την κοινωνική πρόνοια. Το ότι όμως δεν υπάρχει μια παρόμοια κατάσταση σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μας επιτρέπει να κάνουμε κι εμείς μια ισότιμη ανάλυση για όλες τις χώρες. Μολονότι βλέπουμε ότι τα μονογονεϊκά αυτά νοικοκυριά παρουσιάζουν όλο και μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν κάποιες πολιτικές για την υποστήριξή τους, έχουμε όλο και περισσότερα νοικοκυριά τα οποία πλήττονται από την ένδια και την περιθωριοποίηση η κατάσταση των μόνων μητέρων δεν έχει να κάνει μόνο με το ζήτημα της απασχόλησης και της φροντίδας των παιδιών, έχει να κάνει επίσης και με το ότι πολλές φορές ο πατέρας δεν είναι σε θέση να καταβάλει την διατροφή. Όλο και περισσότερο όμως οι μόνες μητέρες αντιμετωπίσουν αυξημένα ποσοστά ανεργίας. Έχουμε και διάφορα ποσοστά ένδυας, φτώχειας, Σύμφωνα με την βάση δεδομένων SILK στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε κάποια ποσοστά όσον αφορά το οικογενειακό καθεστώς ε, των παιδιών εκείνων που ζουν σε νοικοκυριά με μόνους γονείς. Φαίνεται ξεκάθαρο τα παιδιά αυτά κινδυνεύουν περισσότερα από την φτώχεια, από την ένδυα, από όταν ζούσαν σε μια οικογένεια με δύο γονείς. 34% είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος για τα παιδιά εκείνα τα οποία ζουν σε μονογονεϊκές οικογένειες, σε σύγκριση με το 14% κινδύνουν δηλαδή έκθεση στην ένδυα για τα παιδιά εκείνα τα οποία ζουν με δύο γονείς. Και πάλι βλέπουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, το Λουξεμβούργο έχουν ε, τα υψηλότερα ποσοστά έκθεσης δηλαδή στον κίνδυνο της φτώχειας, 44%, μεγάλα ποσοστά παρουσιάζει και η Μάλτα. Στην κεντρική όμως Ευρώπη, βλέπετε εδώ πέρα και τη γραφική παράσταση, στην κεντρική και στην βόρεια Ευρώπη βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια χαμηλότερα ποσοστά, ακριβώς επειδή εκεί υπάρχει ένα πιο έντονο οικογενειακό δίκτυο προστασίας. Και πάλι όμως είπαμε ότι τα επίπεδα της φτώχειας εξαρτώνται από την απασχόληση του γονέα, αν απασχολείται πλήρως ή αν βρίσκεται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης. Σύμφωνα πάλι με τη βάση δεδομένων EU Silk, οι άνεργοι γονεί ή οι γονεί αυτοί οι οποίοι έχουν μερική απασχόληση αντιμετωπίζουν υψηλότερα ποσοστά έκθεση στη φτώχεια. Ο μέσο όρο για τα 25 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 65% όσον αφορά τους άνεργους γονείς, 30% για αυτούς που βρίσκονται σε μερική απασχόληση, ενώ οι μόνοι γονείς που απασχολούνται πλήρως έχουν ένα 15% μόνο ε, κίνδυνο έκθεση ε, φτώχεια. Πάλι θεωρούμε όμως ότι το κοινωνικό και το οικογενειακό δίκτυο μπορεί να προστατεύσει τις μονογενειακές οικογένειες από τον κίνδυνο της φτώχειας και επίσης το θεσμικό πλαίσιο καθώς επίσης και η γενοδορία των κοινωνικών παροχών σε κάθε κράτος μπορεί να βοηθήσει τις οικογένειες αυτές και να τις αποτρέψει από το να εκτεθούν στο κίνδυνο της φτώχειας. Οι μονογενειακές οικογένειες στην Ελλάδα βρίσκονται στο περιθώριο της δημόσιας συζήτησης και της πανεπιστημιακής έρευνας, μόλον ότι αποτελούν πλέον μια ορατή κοινωνική πραγματικότητα. Η έρευνα δείχνει ότι υπάρχει ένας αφανής και λανθάνων παράγοντας στην Ελλάδα για τη δημιουργία τέτοιων μονογονεακών οικογενειών. Τα πρόσφατα χρόνια βλέπουμε ότι οι μονογονεακές οικογένειες αυξάνονται όλο και περισσότερο εξαιτία των αλλαγών που, υφίσταν, που γίνονται στην Ελλάδα στα κλασικά κοινωνιακά πρότυπα και σε κάθε περίπτωση οι μονογονεϊκές οικογένειες στην Ελλάδα αποτελούν μια παραμελημένη ομάδα βλέπουμε ότι ακόμα το θεσμικό πλαίσιο στη χώρα και το κράτος πρόνοιας ακολουθεί ένα παραδοσιακό πρότυπο της οικογένειας, το οποίο είναι παροχημένο, κάπως στατικό. Βλέπουμε ότι ο άντρας εξακολουθεί και θεωρείται ότι είναι ο εργαζόμενος, ο... αυτός ο οποίος ε, ε, φέρνει τα σημαντικότερα έσοδα στην οικογένεια. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υπηρεσίες ε, παιδική μέρημνας και παροχή για τις μενογενειακές οικογένειες, Ακόμα και όταν υπάρχουν υπηρεσίε αυτέ είναι περιορισμένε. Ωστόσο γνωρίζουμε ότι η ιδιότητα του γονέα, η γονική ιδιότητα, αποτελεί ευθύνη τόσο της μητέρας όσο και του πατέρα. Το ότι οι μόνες μητέρες έχουν τη μόνη γονική μέρημνα και την ευθύνη για τη φροντίδα των παιδιών τους τις πρόχνει όλο και περισσότερο στην φτώχεια και δεν τις δίνει πάρα πολλές δυνατότητες να ξεφύγουν από την κατάσταση αυτή. Γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό να εφαρμοστεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα υποστήριξης των μόνων μητέρων βάσει των πραγματικών τους ειδικών αναγκών. Προτεραιότητες θα πρέπει να δοθεί στις δυσκολίες και τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν, το ότι καλούνται να εξορροπήσουν ε, εργασία και γονική μέρημνα, ότι θα πρέπει να τους δίνεται μια ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, κάποιες εξειδικευμένε πολιτικές χρειαζόμαστε επίσης για τις ε, μητέρες, θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν πιο ενεργά στην αγορά εργασίας και να μην συνεχίσει αυτή η νότροπη εξάρτηση από το σύστημα πρόνοιας. Όσον αφορά τώρα τα παιδιά, τα παιδιά των ε, μονογονεκών οικογενειών που έχουν προκύψει από διαζύγιο έχουν ουσιαστικά δύο οικογένειες. Τα παιδιά αυτά καλούνται να αντιμετωπίσουν πολύπλοκα προβλήματα και θα πρέπει να δοθούν σε αυτά εξατομικευμένες λύσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν τι απαραίτητε πολιτικές καθώς επίσης και τα μέτρα κοινωνικής πρόνοιας τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους τις καταστάσει καταστάσεις αυτές που ζουν τα παιδιά αυτά καταλαβαίνετε ότι τα συστήματα κοινωνικής προστασίας πλήττονται από την ε, οικονομική κρίση. Τα συστήματα αυτά στο παρελθόν ε, παίζαν το ρόλο του αυτόματου σταθεροποίητη και βοηθούσαν να μειωθεί η επίπτωση των, ε, της οικονομικής ύφεσης για όλους τους πολίτες, ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες ομάδες. Δεδομένης όμως τώρα της οικονομικής κρίσης, έχει εκτιμηθεί ότι σε ορισμένες χώρες οι κοινωνικές δαπάνες θα αυξηθούν και εξαιτίας οικονομικής κρίσης ορισμένες χώρες ενδεχομένω να μην ανταποκριθούν ανταποκριθούν στι δαπάνε αυτέ. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε ειδικέ πολιτικέ που θα βοηθήσουν του πολίτε εκείνου που βρίσκονται στην πιο δυσμενή θέση. Οι ε, μόνες μητέρε αποτελούν οριακές περιπτώσεις πάρα πολλέ φορές και θα πρέπει να εστιαστούμε στις περιπτώσεις αυτές γιατί συνδυάζουν διάφορα προβλήματα και διλήμματα τα οποία καλούνται τα μοντέρνα σύγχρονα κράτη να αντιμετωπίσουν όσον αφορά στο σύστημα πρόνοιάς του, Θα πρέπει να αναγνωριστούν τα προβλήματα των γυναικών αυτών, καθώ επίση και η μη αμοιβόμενη εργασία που παρέχουν και να καταφέρουν να συνδυάσουμε καλύτερα τόσο τη μη αμοιβόμενη και αμοιβόμενη εργασία των μητέρων αυτών. Ευχαριστούμε, δόκτωρα Λιπράντη, και επειδή διατηρήσατε τον χρόνο ομιλία, Τώρα να δώσουμε το λόγο στην, ε, στα μέλη της Επιτροπής ε, δικαιώματα των γυναικών και ισότητα των φίλων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να δώσουμε το λόγο στην κυρία Γκουρμάη, που είναι μέλος των ε, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι μας δώσατε μια σαφή εικόνα και όπως ξέρετε χρειαζόμαστε περισσότερα στατιστικά στοιχεία για να έχουμε μια σαφή εικόνα. Και ευχαριστώ και την συνάδελφο την κυρία Ματέρα που συντάσσει αυτή την έκθεση γιατί πιστεύω πως η κατάσταση των μητέρων είναι πάρα πολύ σημαντική καθώς η κατάστασή τους είναι δείκτης της κατάστασης της κοινωνίας γενικότερα. Οπότε θα προσπαθήσω να συνοψίσω τις ε, πτυχές που θεωρώ πως πρέπει να συμπεριληφθούν στην έκθεση. Υπάρχουν όλο και περισσότερες ε, αν οι παντρέ μητέρες, αυτό είναι δεδομένο, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, δεν υπάρχει κάποια πολιτική που μπορεί να πάει και να κάνει κάτι τέτοιο. Οπότε, θεωρητική μας βάση πρέπει να είναι η βάση πως όλα τα παιδιά είναι ίσα, ανεξαρτήτως μορφής της οικογένειας στην οποία ζουν και όλες οι μορφές οικογένειών είναι ίσες. Και βεβαίως, ακούσαμε σοκαριστικά νούμερα για ένα 7% των παιδιών που γεννιούνται εκτός γάμου, που σημαίνει πως είναι αρκετά υψηλό το νούμερο. Και βεβαίως η έννοια αυτή της ευθύνης του ενός προς τον άλλον δημιουργεί την έννοια της οικογένειας και όχι η μορφή η ίδια. Τώρα, γιατί χρειάζονται την προσοχή μας οι γονείς που είναι ανήπαντροι, γιατί έχουν τις ίδιες ευθύνε με τα ζευγάρια, αλλά κάνουν τη δουλειά μόνοι τους. Και ευχαριστώ τον συνάδελφο για το ότι κατέστησε σαφές πως ε, στην τελευταία οικονομική κρίση η κατάσταση επιδεινώθηκε. Οπότε οι οικογένειε αυτέ είναι πιο ευάλωτες από άλλες. Θα πρέπει να ξέρουμε πως 91% αυτών των ε, ανήπαντρων γονέων είναι γυναίκε και απειλούνται πολύ περισσότερο από την φτώχεια από ό,τι άλλες οικογένειες και βεβαίως λέμε πως η φτώχεια έχει γυναικείο πρόσωπο και αυτό εξακολουθεί να ισχύει. Πρέπει να αναλύσουμε τα νούμερα, να συγκεντρώσουμε όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω να υπάρχουν περισσότερα δεδομένα προσεχώς. Και βεβαίως θα πρέπει βεβαίως να δούμε πως οι γυναίκες που είναι μόνο τους με ένα παιδί δεν είναι τόσο προετοιμασμένες για τα οικονομικά βάρη και έχουν περισσότερες δυσκολίες στο να μπορέσουν να βρουν οικονομική στήριξη. Και αυτός είναι ο διπλός αγώνας του να είναι κανείς μόνος του σε μια επισφαλή οικονομική κατάσταση με το μόνιμο βάρος βεβαίως της απασχόλησης και τις οικογενειακές ευθύνες και μετά υπάρχει το ζήτημα των συντάξεων και την ανικανότητα αυτών των μητέρων να εξοικονομήσουν χρήματα, να αποταμιεύσουν για τα γεράματα λόγω των οικονομικών βαρών που αντιμετωπίζουν. Επίσης, κάπου άκουσα πως οι μητέρες, οι ανήπαντρες είναι σε χειρότερη κατάσταση από πλευρά υγεία ε, σε σχέση με τι παντρεμένε γυναίκε. Αν αυτό ισχύει, πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Επίσης πρέπει να αναλύσουμε τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτές οι γυναίκες, ειδικά όταν μιλάμε για τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, όπως αναφέρθηκε, και μετά μιλάμε για την απασχόληση γενικώ. Πρέπει να δούμε το ζήτημα της έλλειψης υπηρεσιών, ε, στέγασης, ε, φροντίδας των παιδιών, ε, όχι μόνο τις ώρες γραφείου, αλλά και μετά. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών που τις χρειάζονται αυτές οι οικογένειες απεγνωσμένα από την άλλη για να βοηθήσουμε αυτές τις μητέρες για να συμβιβάσουν οικογενειακή και επαγγελματική ζωή. Πρέπει να ενθαρρύνουμε όλα τα προγράμματα και τις φοροαπαλλαγές ε, και τις ε, παροχές που υπάρχουν από πλευράς ε, εργοδοτών για να δημιουργηθούν χώροι εργασίας φιλικοί προς αυτές τις γυναίκες. Γενικά αυτή η ευπαθή ομάδα θα πρέπει να αποτελέσει στόχο ειδικών κοινωνικών πολιτικών λόγω της υψηλότερη έκθεση της στην φτώχεια και την ανασφάλεια. Οπότε προτείνω να κοιτάξουμε τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη. Και τέλος, κάτι ακόμα το οποίο θεωρώ το πιο σημαντικό. Έχω δει κάποια νούμερα που λένε πως σε κάποιες χώρες η διαχείριση των χρήσεων, δηλαδή η περικοπή των προπολογισμών, πλήττουν χειρότερα τι ανήπαντε μητέρε. π.χ. στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλουμε πραγματικά να πλήξουμε του πιο ευάλωτου. και βεβαίω κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο, να μην δείχνουμε δηλαδή αλληλεγγύη, πρέπει να ζητήσουμε από τις κυβερνήσει να σκεφτούν τον αντίκτυπο που έχουν αυτές οι γυναίκες ή τα παιδιά στο έλλειμμα του προπολογισμού. Δεν πρέπει να φοβόμαστε λοιπόν τον προπολογισμό με βάση το φύλλο. Υπάρχει κάποιο λόγο που ε, έχει κάποιο λόγο που υπάρχει αυτή η έννοια. Και βεβαίως είμαι τυχερή που μετά θα καθίσουμε να τα πούμε με την Μπάρμπαρα πως πριν από λίγο καιρό είχαμε κάποιο σεμινάριο για τους ε, τσάνιπαντες μητέρες στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και ακούστηκε κάτι ενδιαφέρον, προέκυψε εκεί πέρα για το ποια μέτρα βοηθούν ε, αυτού του είδους τα νοικοκυριά και βεβαίως η μεγάλη πλειοψηφία των ανήπαντων γονέων είναι γυναίκες και δεν μπορούν βεβαίως να κρατήσουν και δουλειά και να ε, μείνουν εκτός κοινωνικών παροχών. Να απεξαρτηθούν μάλλον από τις προνοιακές παροχές. Και βέβαια υπάρχει ζήτημα το οποίο δεν αναφέρουμε καθόλου. Π.χ. μια συνάδελφο από την Ολλανδία είχε πει πω οι ανήπαντρε μητέρε στην Ολλανδία εργάζονται περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν και δεν μπορούν να βρουν κάπου να αφήσουν τα παιδιά του. Οπότε είναι σημαντικό να δούμε τι, τι γίνεται. Και βεβαίω υπάρχουν κάποιες χώρες που θα υιοθετήσουν κάποιους στόχους από πλευράς παροχών, αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα, π.χ. Τσεχία, Σλοβακία, Αυστρία και στις λοιπές χώρες. Οπότε νομίζω πως είναι ένα θέμα που είναι επίκαιρο, θα έλεγα, και είμαι σίγουρη πως η Επιτροπή μας και η έκθεση αυτή βρίσκεται σε καλά χέρια γιατί είναι νεαρή συνάδελφος θα συντάξει μια καλή έκθεση και είμαι και στην διάθεσή σας για να βοηθήσουμε γιατί πιστεύω πως είμαστε ίσες, ανήπαντρες ή παντρεμένες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χίλια ευχαριστούμε και σας ευχαριστώ κυρίως για τις ευχές σας. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να κάνει όπως κάνει και όπως πάντοτε έκανε. Και τώρα κυρία Γιανακουδάκη. Thank you, Chair. Um, thank you for... Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Εγώ δεν είμαι σκιώδης συγκήτρια, εκπροσωπώ την ομάδα μου. Αν και είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα και με απασχολεί, γιατί νομίζω μπορεί να είναι κάποιος ε, μόνος γονιός με πολλούς τρόπους, όπως είπαμε. Μου άρεσε ιδιαίτερα η αναφορά που έκαναν και οι δύο μιλήτριες στο ότι μιλάμε για γονείς ανήπαντρους, γιατί είναι 91% γυναίκες αυτή τη στιγμή, αλλά αυξάνονται οι άντρες και θα είναι άδικο στην κοινωνία να μην το λάβουμε αυτό υπόψη όταν εξετάζουμε αυτό το θέμα. Όπως αναφέρθηκε ήδη, είναι ευρύ το φάσμα του τι είναι ένας μόνος γονιός και πώς βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση, π.χ. διαζύγιο. Ο γάμος, όπως είπε μια ομιλήτρια, είναι κάτι το εύθραυστο, να μην πω πως γίνεται κάτι το παλιωμοδίτικο. Και είναι πολύ δύσκολο να επιμείνει κανείς καμιά φορά. Έχουμε χείρες, διαζύγια, γονείς εκτός γάμου, εκτός ας πούμε της ε, κανονικής κατάστασης. Οπότε αυτό επηρεάζει την κατάστασή τους και τη θέση τους και ίσως να μην είναι σε τόσο ισχυρή θέση όσο θα ήταν γιατί κάποιος ο οποίος έχει μια οικονομική άνεση και έχει βοήθεια των γονιών ε, ή είναι χείρα θα είναι σε κάπως καλύτερη κατάσταση σε σχέση με κάποια η οποία είναι μόνη μητέρα και έχει εξοριστεί εντό εικόνων από του γονεί τη και την κοινωνικό τη περίγυρο κτλ. Οπότε ας δούμε τι μπορεί να γίνει. Μέχρι στιγμή πολλοί είπαν ε, για οικονομική βοήθεια ναι. Οικονομική βοήθεια πάντα καλό πράγμα είναι. Στο Ηνωμένο Βασίλειο εμείς ε, εξετάζουμε το εισόδημα όσων είναι μόνοι τους, έχουμε επίδομα παιδιών, έχουμε διάφορους τρόπους να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Τώρα, για προϋπολογισμό, ειδικά για τα φύλλα, δεν είμαι τόσο σίγουρο, γιατί όταν μιλάμε για προϋπολογισμό για τα φύλλα για συγκεκριμένες ομάδες, π.χ. μπορούμε να μιλήσουμε και για προπολογισμό για εθνικές μειονότητες, για ανάπηρους. Υπάρχουν διάφοροι τομείς που χρειάζονται ξεχωριστό προπολογισμό και στο τέλος θα απομείνει ένα ελάχιστο ποσοστό πληθυσμού που δεν θα έχει φοροαπαλλαγές και δεν θα υπάρχουν χρήματα. Οπότε εγώ εξετάζω την ευρύτερη εικόνα πέρα από την άμεση οικονομική στήριξη και έχει πρόσβαση στις πληροφορίες και στο τι προσφέρεται. Εγώ θα πάω στην παλιά αυτή φράση που έχει ξαναέρθει στη μόδα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την λεγόμενη μεγάλη κοινωνία που ανέφερε ο Πρωθυπουργό μας. Ε, εκεί πέρα αναλαμβάνει η κοινωνία την ευθύνη και βοηθάει πολύ περισσότερο. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσω ομάδων που θα βοηθούν, θα μοιράζονται εμπειρία για τη φροντίδα των παιδιών, αλλά σε πιο εθελοντική βάση. Η Ελλάδα είναι ένα καλό παράδειγμα αποκλεισμού των ε, μονογονεϊκών. Καλά, προφανώς αν είναι κανείς χείρα δεν αποκλείεται. Αν είναι χωρισμένη, ίσως όχι τόσο τώρα πια, αλλά αν υπάρχει παιδί εκτός γάμου, ε, είσαι αποκλεισμένη από ό,τι ξέρω την ελληνική κοινωνία. Στην Αγγλία, ίσως να είναι κάπως πιο ανοιχτόμυαλη η προσέγγιση, συνοψίζοντας. Υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να δούμε, να δούμε τα εύκολα προβλήματα, τα οικονομικά, τα την άμεση στήριξη, την οικονομική, αλλά και τα πιο δύσκολα, τα έμεσα ζητήματα, δηλαδή τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, το παιδί που δεν αναφέρθηκε καθόλου, τι συμβαίνει σε αυτά τα παιδιά, εάν προέρχονται από κάποιο ασταθές περιβάλλον, γιατί αν μια μητέρα προσπαθεί να ανατρέψει παιδί χωρίς τη στήριξη της οικογένειάς της επηρεάζεται το παιδί. Οπότε η προσέγγιση μου είναι να λάβουν υπόψη την προσέγγιση της μεγάλης κοινωνίας στα κράτη-μέλη, να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να συνεργαστούν, να αποδεχτούν αυτούς τους γονείς και να τους βοηθήσουν όπου μπορούν. Ευχαριστούμε κυρία Γιανακουδάκη. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συνεισφέρει και εκείνη στο θέμα, η Μαρία Αν από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Όχι λάθος, άλλη συνάδελφος ακόμα. Υπάρχουν και άλλες συνάδελφοι που θέλουν να παρέμβουν. Ας ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα και μετά τις υπόλοιπες συναδέλφους που θέλουν το λόγο. Uh, Ευχαριστώ που προσκαλέσατε την Κομισιόν να λάβει μέρος σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ προσωπικά έχω εμπλακεί στα ζητήματα που αφορούν τους γονείς ασχολούμαι με αυτά τα ζητήματα εδώ και 16 χρόνια. Πρώτα απ' όλα δούλευα στη μονάδα ισότητας των φίλων και εδώ και 7 χρόνια με τη μονάδα που ασχολείται με την κοινωνική ένταξη και μαζί με την κυρία Τριφιλέτη ασχολούμαστε με αυτή τη μελέτη για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα να τονίσω το ζήτημα των τρόπων που οδηγούν στο να είναι κανείς μόνος γονιός. Όπως είπε η κυρία Γιανακουδάκη, ειδικά σε κάποιες χώρες, ο δρόμος με τον οποίο καταλήγει κάποιος στο να είναι μόνος γονιός είναι καθοριστικός για το πώς τον αντιμετωπίζει η κοινωνία. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο αναφέρθηκε και είναι προέκυψε από την έρευνα της κυρίας Τριφυλέτη είναι πως το ποσοστό δραστηριοποίησης ε, των γυναικών που είναι μόνες τους ε, ποικίλει πάρα πολύ ανάλογα με τη στήριξη που έχουν από το κράτος ε, πρόνοιας. Γιατί στις νότιες χώρες κινητοποιούνται πάρα πολύ περισσότερο γιατί το κράτος πρόνοιας δεν έχει επιδόματα σε μετρητά ή άλλα επιδόματα για να βοηθήσει τις ανήπαντρες μητέρες. Ένα τρίτο ζήτημα, το οποίο θα ήθελα να αναφέρω, είναι πως μέχρι στιγμής το μοντέλο συμβιβασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής βασίζεται στο, στην υπόθεση πως υπάρχουν δύο εργαζόμενοι και δύο γονεί στον οικοκυριό. Και εκεί πέρα βεβαίω υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν για να λάβουμε υπόψη τον αυξανόμενο αριθμό μόνο γονεϊκών οικογενειών. Ένα άλλο θέμα το οποίο αναφέρθηκε ήταν αυτό του ότι θα πρέπει να θεωρείται μεταβατική φάση στην ζωή ενός ατόμου το να είναι ανήπαντρος γονιός και άρα το κράτος πρόνοιας θα πρέπει να κληθεί να συνεισφέρει περισσότερο από ό,τι συνήθως. Και να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να φύγουν από αυτή η κατάσταση. Παραδείγματο χάρη, θα έλεγα να σκεφτούμε πρωτοβουλίες όπως αυτή που υπάρχει στη Γαλλία, το εισόδημα Ενεργού στήριξη, ενεργού αλληλεγγύη για αυτούς που παίρνουν επίδομα ανεργίας και για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα έξοδα εάν βρουν μια νέα δουλειά παραδείγματο χάρη, π.χ. τη φροντίδα του παιδιού ή τα τη μεταφορά, να έχουν ένα έξτρα εισόδημα. Και άρα το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και για γονιούς ε, μόνους που αρχίζουν να δουλεύουν. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες πρακτικές που προκύπτουν σε πολλές χώρες ε, όσον αφορά την στήριξη στην ανατροφή των παιδιών. Υπάρχουν όλο και περισσότερες ομάδες που συστήνονται για να δώσουν ε, στήριξη στους γονείς και βεβαίως αυτή είναι μια πρωτοβουλία που καλό θα ήταν να προωθηθεί. Τώρα όσον αφορά την πολιτική. Όπως ξέρετε, από το Δεκέμβριο του 2010 έχουμε την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στο πλαίσιο αυτό έχουμε δύο προτεραιότητες υπό τις οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως προτεραιότητα οι ανυπαντρές μητέρες. Πρώτα απ' όλα, στο πλαίσιο της παιδικής φτώχειας βασικός τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την φτώχεια των παιδιών είναι μέσω της στήριξης των γονιών, των Και υπ' αυτή την έννοια μια μεγαλύτερη στήριξη στους ανήπαντρους γονείς θα ήταν κάτι το θετικό, κυρίως γιατί όπως αναφέρθηκε σε ορισμένες χώρες υπάρχει στίγμα για του ανήπαντρους γονεί και αυτό έχει συνέπειε για τα παιδιά. Ενώ εάν έχουμε παροχέ για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως του καθεστώτος των γονιών, τότε ε, αυτό θα βοηθήσει του πάντες. Μετά, ο δεύτερο τομέα στον οποίο θα μπορούσαμε να παρέμβουμε, είναι η νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων που καλύπτει τα έτη 2010 με 2015 εκεί υπό το θέμα του χάσματος του εισοδήματος των δύο φίλων μπορούσαμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα συγκεκριμένα προβλήματα που ε, αντιμετωπίζουν οι ανήπαντρες μητέρες λόγω της έλλειψης επαρκούς εισοδήματος λόγω διαφόρων ζητημάτων και εμποδίων που αντιμετωπίζουν και αναφέρθηκαν ήδη. Αυτά για την ώρα και ίσως να επανέλθω αργότερα με συγκεκριμένες προτάσεις που προέκυψαν στη διάρκεια των ετών, σε σεμινάρια και άλλα φορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Επιτροπή για τη δική της συνεισφορά. Επιφυλασσόμεθα να ξαναζητήσουμε τη δική σας άποψη. Και τώρα για μια σύντομη παρέμβαση Ιδίω αν θέλετε να απευθύνετε ερωτήματα προ τι εμπειρογνώμονε. Σύντομα παρακαλώ. Η κυρία Τόμψον για του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να πω πως θέλω να ευχαριστήσω τις ομιλήτριες για τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και είμαι και εγώ βεβαίω στην ομάδα αυτή των εμπειρογνωμόνων, καθώς έχω ήδη άπειρα για το να είναι κανείς μόνη μητέρα. Και είπατε πράγματα για την περισσότερη έρευνα και συμφωνώ για την πολυπλοκότητα του μοτίβου που παρουσιάζεται σε διάφορες χώρες, αλλά ένας καθοριστικός παράγοντος, στη δική μου εμπειρία τουλάχιστον, είναι όταν συγκρίνουμε, είναι να δούμε πόσα παιδιά έχει κανείς και όταν μιλάμε για μητέρες της ε, ε, χώρες του Νότου που είναι πιο δραστήριες. Ναι, γιατί έχουν ένα παιδί, ενώ στις βόρειες χώρες έχουν δύο ή περισσότερα. Και εγώ θεωρώ πως μία μητέρα μόνη της με ένα παιδί έχει περισσότερες δυνατότητες για καριέρα από μία παντρεμένη μητέρα με τρία παιδιά και άντρα, γιατί δεν έχει μόνο τα τρία παιδιά, έχει και τη δουλειά της νοικοκυριάς, της συζύγου. Και βεβαίω ε, τα παιδιά πρέπει και αυτά να εκπαιδευτούν και υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντε που ορίζουν το πώ ε, ε, είναι η κατάσταση του καθενό στην κοινωνία. Μια πρακτική εμπειρία που έχω από τη χώρα μου, τη Δανία, είναι πως, από ό,τι έχω δει σε ευρωπαϊκές χώρες, τα λεφτά, η συνεισφορά από τους πατεράδες στις μητέρες δεν είναι ζήτημα μεταξύ των γονιών, είναι ζήτημα μεταξύ του πατέρα και του κράτους και του κράτους και της μητέρας μετά. Οπότε το κράτος δίνει τα λεφτά στη μητέρα κάθε μήνα ή όποτε τέλος πάντων τα έχουν κανονίσει και μετά ο πατέρας πρέπει να πληρώσει το κράτος. Εάν ο πατέρας δεν μπορεί να πληρώσει, τότε είναι θέμα δικό του και του κράτους. Και μόλις βρει δουλειά, το κράτος θα πάρει τα λεφτά από το μισθό του απευθείας. Και έχω δει στην Πορτογαλία, π.χ. σε άλλε χώρε, οι μητέρε να μην λαμβάνουν αυτά τα λεφτά και να είναι φοβερά φτωχέ. Εάν κάνουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία ως προς αυτό, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, ε, το θέμα της εκπαίδευσης. Η Μάλτα και η Ιρλανδία έχουν πάρα πολλές ε, έφηβες μητέρες γιατί δεν έχουν πρόσβαση στην ε, άμβλωση και πηγαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί γίνεται τώρα αυτό. Τώρα στη χώρα μου υπάρχει μια τάση να έχουμε όλο και περισσότερα παραδείγματα ε, εφήβων μητέρων. Ταυτόχρονα βλέπουμε τα τελευταία 10-15 χρόνια πως η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση έχει χαμηλή προτεραιότητα, οπότε δεν έχουν τη γνώση και βλέπω πως ε, θεωρούν οι γυναίκες πως είναι εναλλακτική καριέρα το να γίνουν μια νεαρή μητέρα και να ζήσουν από τα επιδόματα αν δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Οπότε και αυτό είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα και πρέπει να το ερευνήσουμε αυτό το θέμα των έφηβων μητέρων γιατί είναι πολύ κακή αφετηρία για τα παιδιά. Οπότε βλέπω εγώ με την πλειοψηφία των μητέρων να είναι τελείως ανίκανες στα 16 τους να φροντίσουν δύο-τρία παιδιά που κάνουν. Αυτή ήταν η δική μου συνεισφορά. Ευχαριστούμε κυρία Τόμσον. Και τώρα η κυρία Κώστα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την εισηγητρία βρίσκονται το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Όλε λοιπόν θα συμβάλλουμε στη συζήτηση και υπό το φω αυτών των πολύ ενδιαφερουσών ε, παρουσιάσεων. Νομίζω ότι συγκλίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό μας εξυπηρετεί, διότι μπορούμε έτσι να αντιμετωπίσουμε σημαντικά φαινόμενα χάρη στη δική σας τη συμβολή. Κατά πρώτον, νομίζω πρέπει να επεξεργαστούμε ορισμένα συγκεκριμένα σημεία και να κάνουμε και κάποιε συστάσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά πρώτον, όπω είπαν κάποιοι συνάδελφοι, υπάρχει μεγαλύτερη στατιστική σύγκληση, δηλαδή εμβάθυνση, μελέτη ε, ε, στην πράξη και περισσότερη ε, οριζόντια μελέτη των φαινομένων και των, του τι συμβαίνει στο επίπεδο της ηλεκτρονική πρόνοια. Όλα αυτά χρειάζονται και καθώ και εναρμόνιση των παραμέτρων. Εσεί μιλήσατε ε, για την ε, Γαλλία, για τα εξαρτώμενα ε, παιδιά. Τα εξαρτώμενα τέκνα που σε κάποιε χώρες ορίζονται, σε κάποιες άλλες όχι, η κατάσταση διαφέρει. Επίσης, ε, οι παράμετροι του κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας, τα δίκτυα, τα άτυπα, τα επίσημα, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε με περισσότερη ακρίβεια. Και θα ήταν πολύ καλό και η δική μας Επιτροπή να δώσει μια όθηση σε αυτό το είδος την έρευνα. Να, να συμμετέχουμε και εμείς σε μια τέτοια μελέτη σύγκλησης. Κατά δεύτερον, μιλώ τώρα περισσότερο θεωρητικά και μετά θα μιλήσω κατά πολιτικά ζητήματα, νομίζω ότι χρειαζόμαστε δεδομένα τα οποία να μην είναι τόσο προβληματικά. Υπάρχουν μεγαλύτερε αποκλήσεις. Δεν θέλω να πω ότι υπάρχουν δύο ευρώ. δύο Ευρώπες, αν και σε έναν βαθμό αυτό ισχύει, αλλά Υπάρχουν ε, δύο διαφορετικές ιστορίες, ιστορικές παραδόσεις στην Ευρώπη, στο Βορρά. Έχουμε κυρίως μητέρες ανήπαντρες ε, με μικρά παιδιά. Οι πατέρες είναι πολλές φορές φοιτητές με μια προσωρινή εργασία, είναι για εκείνη πιο αδύναμη. Υπάρχει μια τέτοια πολιτιστική παράδοση στις χώρες αυτές. Η πρώιμη μητρότητα όμω δεν αντιμετωπίζεται τόσο απλά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η εγκυμοσύνη είναι πρόσβαση, είναι πρόσβαση στην ε, κοινωνική πρόνοια. Ε, γιατί βλέπουμε να ισχύει το ίδιο φαινόμενο και σε χώρε που δεν έχουν τέτοια κοινωνική πρόνοια. Υπάρχει επιθυμία για μητρότητα εκεί. Ε, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την συμβουλευτική μα, τι αποκρίσει μπορούμε να δώσουμε κάπω πιο οργανωμένε, διαδεδομένε. Ε, ένα δεύτερο ζήτημα που προκύπτει είναι μεγάλη αύξηση 37% που όμως υποκρύπτει δύο πολύ διαφορετικές ε, πραγματικότητες. Περισσότερες νέες ε, και ανήπαντρες στο βορρά, περισσότερα διαζύγια και μονογονικές οικογένειες στο νότο. Εδώ θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη μελέτη για τα παιδιά που είναι γεννημένα εκτό γάμου και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να μειώσουμε τα δικά του τα δικαιώματα. Πρέπει να προστατεύονται κατά τον ίδιο ακριβώ τρόπο με τι γυναίκε και τα παιδιά που έχουν ε, βγει από ένα διαζύγιο. α, το σε τι κατάσταση βρίσκονται τα παιδιά σε σχέση με του γονεί είναι ένα θεμελιώδη στοιχείο που πρέπει να ξεκινήσουμε. Από την άλλη όμω είναι αναγκαίο να αναζητήσουμε έναν συνδυασμό πολιτικών που να προσαρμόζονται στι ανάγκε των διαφορετικών μορφών οικογενειών, ανάλογα με το αν είναι ο πατέρα ή η μητέρα μόνη και τι καταστάσει αντιμετωπίζουν. Και θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω με αυτά. Εσείς μας δώσατε πολλές πληροφορίες, ε, προέκυψαν κάποια στοιχεία ενδιαφέροντα. Με ενδιαφέρει πολύ αυτό που είπε ο συνάδελφο Τόμσον. Νομίζω ότι είναι καθοριστική σημασία. Το κράτο να λειτουργεί ω εγγυητή κατά κάποιο τρόπο σε περιπτώσει διαζυγίου λόγου χάρη. Εκείνος να, εκείνο να δίνει τη διατροφή. Ακόμη και όταν ο πατέρα δεν είναι σε θέση, όχι μόνο άμα δεν θέλει, εδώ λοιπόν ίσως θα μπορούσε να υπάρχει μια πρόταση εναρμόνησης του τι γίνεται στην Ευρώπη. Και οι ερευνήτριές μας νομίζω ότι συνεισέφεραν σε αυτή την ιδέα σε σχέση με, την, με το policy mix που υπάρχει στην Ευρώπη. Κατά τη δική σας άποψη υπάρχουν μοντέλα ή διαφορετικοί τύποι παρέμβασης ή μπορεί κάθε χώρα ανάλογα με την ιστορία της, την παρουσιασή της να συνεχίζει την παρέμβασή της ε, στο πλαίσιο αυτών των συνδυασμένων πολιτικών βλέπουμε ότι τα ανεπίσημα δίκτυα, οι μεγαλύτερε οικογένειε στο Νότο έχουν κρατήσει περισσότερο, είναι μακροβιότερε. Ενώ στο Βορρά φέρεται να υπάρχει περισσότερη τάση προ την εδραίωση των κρατικών πολιτικών. Άρα, φαίνεται να υπάρχουν δυνατότητε, πόροι, ε, οικογενειακά δίκτυα, άτυπη κοινωνική πρόνοια, πέραν τη επίσημη κρατική παρέμβαση. Και αυτά θα μπορούσαν να αποτελούν μέρο του συστήματο. Νομίζω ότι θα, μας, θα ακούσουμε και άλλα σήμερα για τέτοιες ευέλικτες υπηρεσίες, αλλά και η οργάνωση της επαγγελματική ε, ε πρέπει να είναι πιο ευέλικτη. Θα πρέπει να έχουμε καλύτερη αναγνώριση των διαφορετικών τύπων οικογενειών, αλλά και διαφορετικές πολιτικές με αναγνώριση της αλληλοβοήθειας και τα σχετικά δίκτυα και το αναγνώριση του γεγονότο ότι μπορεί η μονογονεϊκή οικογένεια να είναι μια προσωρινή φάση τη ζωή του γονέα. Δεν είναι κάτι απαραίτητα μόνιμο. Σήμερα το πανόραμα αυτό τη Ευρώπη μα δείχνει λύσει πολύ ενδιαφέρουσε, τι οποίε θα μπορούσαμε να επεξεργαστούμε μαζί με την εισηγήτρια για να ευνοήσουμε αυτήν την ισχυρή συμβολή του Ευρωκοινοβουλίου. Ευχαριστούμε, κυρία Κώστα. Και τώρα να δώσουμε σύντομα το λόγο στι εμπειρογνωμονέ μα για να ολοκληρώσουμε. Έχουμε μια πρώτη κατεύθυνση μας που τα μέλη της Επιτροπής μας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ας κινηθούμε λοιπόν σε αυτή την πορεία. Έχετε πέντε λεπτά περίπου. Σε πέντε λεπτά είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω. Τέθηκαν όμως πολλές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και ήθελα να αποσαφηνίσω κάποια πράγματα τα οποία τα είπα πολύ εντάχει. Νομίζω ότι επανέρχεται αυτή η πρόταση που σχεδόν έχει ήδη διατυπωθεί. Η Ευρώπη να αναλάβει την ευθύνη, να δώσει κατεύθυνση στις πολιτικές της τέτοια, που να περάσουμε και σε μια πολιτιστική καμπή, μια καμπή στην νοοτροπία μας. Μια γυναίκα πολύ νέα που δεν έχει ακόμη δουλέψει, δεν έχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Και να θέλει δεν μπορεί να πληρώσει την... τα έξοδα του διαζυγίου. Και ένας πατέρας το ίδιο. Και επίση υπάρχουν και κοινωνικέ πραγματικότητε καινούργιε εξαιτία αυτής τη συλλογική μεταβολή των οικογενειακών ε, σχηματισμών. Θα πρέπει λοιπόν να τι αναγνωρίσουμε όπως έχουν, χωρί να στιγματίζουμε κανέναν. Είδαμε και δύο παρεμβάσει να συγκλίνουν στο εξή, αλλά το κράτο δεν είναι ακριβώς ο εγγυητή του ποσού που ουσιαστικά καταπολεμάται και συμπληρώνει το τη διαφορά της μόνης μητέρας από το όριο της φτώχειας. Όπως μας λέει το αγγλικό μοντέλο για τον ε, πατέρα που δεν είναι σε θέση. Ίσως υπάρχει και ένας ε, νέος τύπος φτώχειας που θα έπρεπε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε. Και κάτι άλλο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι ακριβώς, αλλά ίσως το είπα και προηγουμένως, χωρίς να έχω το χρόνο να το αναλύσω, νομίζω ότι πράγματι οι χώρες που ακριβώς είχαν πρόωρα τέτοια φαινόμενα μπόρεσαν να προσαρμοστούν αρκετά. Κάποιοι άλλοι όμως δεν έχουν οικογενειακή πολιτική και δεν σκοπεύουν να έχουν τέτοια, ειδικά με συνέπεια. Νομίζω πολύ σημαντικό είναι τα μέτρα να, που αφορούν τις, μονογονικές οικογένειες να στοχεύουν στις χώρες όπου υπάρχουν ήδη οικογενειακές πολιτικές να υπάρχει καλός συνδυασμός, συντονισμός με τα όσα ήδη προβλέπονται. Και επίσης στις χώρες όπου αυτό δεν προβλέπεται, τουλάχιστον η κοινωνική προστασία, η πρόνοια να κάνει πρόληψη για τα ζητήματα αυτά. Κάποιες φορές υπάρχουν απλώς θεωρητικές κατηγορίες στα πλαίσια της κοινωνικής προστασίας, αλλά δεν υπάρχει δημόσια αναγνώριση ότι υπάρχει αυτή η κοινωνική πολιτιστική μεταβολή σε επίπεδο κράτου. Και το να έχει κανείς παιδιά εκπροσωπεί και ένα κόστος. Όλα αυτά λοιπόν σίγουρα αποτελούν μέρος μιας νέας κατεύθυνσης. Η ευρωπαϊκή πολιτική, η κοινωνική πρόνοια πρέπει να οδεύσει σε μια συγκεκριμένο προορισμό. μειώνεται πάρα πολύ το ποσοστό γεννήσεων στις ε, χώρες της Ευρώπης. Έτσι μου φαίνεται σημαντικό και σε επίπεδο συστάσεων όλα αυτά τα θέματα να συζητηθούν και δημοσίως. Ώστε να υπάρξει μια συνολική ζήμωση. Θα μπορούσαμε μάλιστα να φανταστούμε και πολιτικές με μηδενικό κόστος που ωστόσο να αναγνωρίζουν τρόπον την άτη συμβολή των μονογονεϊκών οικογενειών. Η στήριξη των δικτύων αλληλοβοήθειας των ατύπων είναι και αυτό ένα τέτοιο στοιχείο. αλλά και η διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες childcare για τους μόνους γονείς. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι οι ανήπαντρες μητέρες Κάποιε φορές έχουν προτεραιότητα στην πρόσβαση. Αλλά χρειάζεται και κοινωνική αναγνώριση. Δηλαδή, από τη μια έχουμε τι δείξει του ίδιου νομίσματο. Από τη μια ε, αναγνωρίζεται η προτεραιότητα πρόσβασή του, από την άλλη έχουν στιγματιστεί. Σα το λέω και σα βλέπω ε, να εκπλήσεστε. Αλλά Υπάρχουν σε πολλέ χώρε αυτά τα προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν να συμβάλλουμε στην αλλαγή νοοτροπία, τάση, την πολιτιστική αλλαγή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θα γίνει πολύ δύσκολο αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα. Ε, ευχαριστούμε την κυρία Τρεφιλέτη για την ε, συμβολή τη και τώρα να δώσουμε το λόγο στην δόκτωρα Αλιπαράντη. Θα μιλήσω ελληνικά. Υπάρχει διερμηνία τα προβλήματα όπως είδαμε και όπως τονίστηκαν από όλες τις ομιλήτριες και από τις, ε, ε, τα μέλη της Επιτροπής ΦΑΜ είναι πάρα πολλά και συνδέονται τόσο με τους γονείς όσο και με τα παιδιά αυτά τα οποία έχουν διαφορετικά προβλήματα ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση της μητέρας ή του πατέρα. Επίσης ελέγχθηκε ότι θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται και με τον μόνο πατέρα. Δηλαδή δεν θα πρέπει μόνο να επικεντρωθούμε στα προβλήματα των μόνων μητέρων. Έχει αρχίσει και η μορφή οικογένειας με μόνο πατέρα, ιδίως στη Σουηδία είναι σε μεγαλύτερο βαθμό, να αρχίσει και αυτό το να υπάρχει. Είναι υπαρκτή. Από ό,τι είδα κάτι στατιστικές, 26% των μόνων γονέων στην Σουηδία είναι πατέρες. Οπότε θα πρέπει να ληφθούν όλα αυτά τα προβλήματα υπόψη από τις ε, χώρες ώστε να δημιουργηθεί ε, μια ε, ισχυρή, ένα επίπεδο αντιμετώπισης αλλά διαφοροποιημένο. Επίσης ελέγχθη ότι στις μεσογειακές χώρες υπάρχουν τα, έχουν παραμείνει τα οικογενειακοί δεσμοί και έχουμε λοιπόν αρκετά οικογενειακά δίκτυα που συχνά υποκαθιστούν το κράτος πρόνοιας. Αυτά σιγά σιγά βέβαια και σε αυτές τις χώρες τις μεσογειακές και από την εμπειρία μου αρχίζουν να εξαστερούν. Δεν μπορούμε δηλαδή να επαναπαυθούμε μόνο στα κοινωνικά δίκτυα ούτε στις εθελοντικές οργανώσεις. Ελέγχθηκε ότι στην Αγγλία είναι η κοινωνία, η ανοιχτή κοινωνία που θα μπορέσει να υποκαθαστήσει το κράτος πρόνοιας. Δεν ξέρω αν μπορεί αυτό να εφαρμοστεί σε όλες τις κοινωνίες. Ε, και νομίζω ότι ε, η κοινωνία των πολιτών έχει αναπτυχθεί για άλλες παρεμβάσεις ε, και συχνά είναι πολύτιμη η κοινωνία των πολιτών, αλλά σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας, όπως έχει αποδειχθεί, δεν είναι τόσο αποτελεσματική η παρέμβαση. Τουλάχιστον στις χώρες μεσογειακές, που δεν υπάρχει τόσο αναπτυγμένη η κοινωνία των πολιτών. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστούν όλες οι πτυχές της μονογονεϊκότητας, της μόνης, ε, του μόνο, των μόνων γονέων, ανεξάρτητα από το φύλλο του, γονέα, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των γυναικών και των παιδιών που όπως ελέγχθη είναι διαφορετικά και διαφοροποιούνται ανάλογα αν είναι η μητέρα χωρισμένη, αν είναι ε, χείρα, αν είναι ανήπαντρη. Οπωσδήποτε η μονογονικότητα δεν είναι μια, ε, δεν είσαι φόρου ζωής μόνος γονέας, αλλάζει, ε, μπορεί να είσαι μόνος γονέας, να, να, να κάνεις παιδί μόνη, μετά να παντρευτείς τον σύντροφό σου, αλλά οπωσδήποτε και η παρουσία και των δύο γονέων είναι πολύ σημαντική. Ελέγχθηκε για τις ε, ανήλικες μητέρες ότι έχει αρχίσει μια τάση στην Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες ε, νομίζω ότι οι ευθύνες και των γονέων της ανήλικης μητέρας πρέπει και αυτοί να αναλάβουν κάποιες ευθύνες. Δεν μπορεί το κράτος όλα να τα αναλάβει. Θα πρέπει και οι σύντροφοι και οι πατέρες και οι πατέρες των ανήλικων μητέρων να έχουν και αυτοί ε, να ευαισθητοποιηθούν ώστε όχι ότι κάνω ένα παιδί, το αφήνω σε μια γυναίκα και τέρμα. Να υπάρχει δηλαδή μια συμβολή και από αυτή τη μεριά. Ε, και θεωρώ ότι θα, δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει μια, ε, μια σφαιρικότερη αντιμετώπιση από το κράτος, από την κοινωνία των πολιτών και γενικότερη αντιμετώπιση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί πραγματικά στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία πολιτική που να απευθύνεται μόνο για τις μόνες μητέρες. Υπάρχει για τις μητέρες που τα παιδιά τους είναι σε κρίσεις, για φτωχές, για αυτά, αλλά για ανήπατρες δεν υπάρχει και μπαίνουν, παίρνουν κάποιον πάρα πολύ μικρά επιδόματα με αυτές τις γυναίκες τις αγκαταλελειμμένες που τις έχει καταλήψει ο πατέρας ή που είναι στη φυλακή ο πατέρας και δεν μπορεί να πληρώσει ή διάφορες τέτοιες καταστάσεις χωρίς να απευθύνονται ε, μόνο στις ανήπαντρες μητέρες ή στις μόνες μητέρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία, την ε, δόκτωρα Λιπράντη. Και τώρα περνάμε στη δεύτερη ομάδα προσκεκλημένων, στο δεύτερο πάνελ. Θα μπούμε στην ουσία του ζήτηματο που σήμερα συζητούμε. τι ανήπαντρε μητέρε, single mother. Ευχαριστώ ιδιαίτερω τι εμπειρογνώμονε που ήδη παρενέβησαν. Και τώρα προσκαλώ τις υπόλοιπε εμπειρογνωμονε του δεύτερου πάνελ, την πρόεδρο του MME, ε, την κυρία Λίντεκερκ, και την εκπρόσωπο των μόνων μητέρων, sí. του δικτύου μόνων μητέρων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 να είναι και πολύ συγκεκριμένη και αποδοτική. E και τώρα καλώ την πρόεδρο, την πρόεδρο του ε, Διεθνούς Κινήματος ε, των Μητέρων. Είναι μια κυβερνητική οργάνωση που έχει ιδρυθεί από το 1947 και θέλει να δώσει έμφαση στο όρο των μητέρων στο πλαίσιο των κοινωνιών ε, και βεβαίως και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ σύντομα ε, να χαιρετήσω και τη Γενική Γραμματεία του κινήματος αυτού, την Καρολίνη Μπομασέη που βρίσκεται μαζί μας. Τώρα θα δώσω το λόγο στην πρόεδρο του κινήματος αυτού. Με συγχωρείτε, ε, να θυμίσω απλώς ότι έχετε 15 λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρία Ματέρα. Θα μιλήσω στα γαλλικά. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα να πάρω το λόγο στην Επιτροπή σας και να εκπροσωπήσω όλες αυτές τις μητέρες οι οποίες βρίσκονται σε δινή θέση. Θα ήθελα να είμαι επίσης συγκεκριμένη και σύντομη στις συστάσεις που θα κάνω, ορισμένες από τις οποίες βέβαια ήδη αναφέραμε, ήδη ανέφεραν οι προαλήσασες. Όπως είπε η κυρία Ματέρα, το Παγκόσμιο Κίνημα για τις Μητέρες είναι μη κυβερνητική οργάνωση που δεν ακολουθεί κάποια πολιτική κατεύθυνση και που έχει συμβουλευτικό ρόλο στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Θέλουμε να προωθήσουμε το ρόλο της μητέρας στα πλαίσια της κοινωνίας και δίπλα στις διεθνείς και εθνικές δομές και θεσμικά όργανα. Βρισκόμαστε επί τόπου προκειμένου να ακούμε περισσότερο τις ημέρες και βρισκόμαστε για αυτό το λόγο εδώ σήμερα προκειμένου να καταφέρουμε να μεταφέρουμε σε εσά την φωνή των γυναικών αυτών που μέσω των εκλογών εσείς εκπροσωπείτε. Είναι γυναίκες και μητέρες και ουσιαστικά περισσότερες βρίσκονται στη θέση την οποία εξετάζετε εσείς σήμερα. Δηλαδή είναι μόνες γυναίκες, μητέρες. Ήδη από το 1947 η οργάνωσή μου προσπαθεί να προωθήσει τον πολύ σημαντικό κοινωνικό ρόλο που μπορούν να δραματίσουν οι γυναίκες μέσω της μητρότητας παγκοσμίω. Γι' αυτό το λόγο η MMM Ευρώπης συνεργάζεται σε ένα σχέδιο της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να δημιουργηθεί το Family Platform, αυτή η πλατφόρμα οικογενειακή η οποία θα ολοκληρωθεί το 2011 και στόχος της είναι να δημιουργηθεί απαραίτητη βάση προκειμένου να χαραχθεί μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τις οικογένειες. Πρόκειται για μια εργασία στην οποία θα κληθείτε εσείς να συμβάλλετε, κυρίες και κύριοι βουλευτές και για την εργασία αυτή θα θέλαμε και εμείς να συμβάλλουμε με τη δική μας εμπειρογνωμοσύνη. Στα πλαίσια αυτού του Family Platform, η MMM Ευρώπης ανέλαβε ως καθήκον να συντάξει μία έκθεση για την κατάσταση των μητέρων στην Ευρώπη, προκειμένου να συνταχθεί η έκθεση αυτή και προκειμένου να καταφέρουμε πραγματικά να εκπροσωπήσουμε τις μητέρες και να μιλάμε αντί για αυτές. Κάναμε μία online έρευνα όπου 11.000 περίπου μητέρες στην Ευρώπη συμμετείχανε. Η έρευνα αυτή έγινε από το Φεβρουάριο μέχρι τον Αύγουστο του 2010 σε 16 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 10 γλώσσες. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ σήμερα που θα είμαι σε θέση να μιλήσω εξ ονόματος των μητέρων αυτών, βασιζόμενοι σε αυτή την έρευνα. Από τις 11.000 μητέρες που συμμετείχανε 1500 ε, ανήκουν σε μονογονεακές οικογένειες και μας μίλησαν για τις βασικές τους προτεραιότητες. Οι περισσότερες ε, είναι διαζευγμένες ή χωρισμένες. Μία στις τέσσερις μας είπε ότι δεν παντρεύτηκε ποτέ και δεν έχει συζήσει και περίπου μία στις δέκα είναι χείρα. Δεν λάβαμε απαντήσεις από τις μόνες μητέρες κάτω από 18 ετών. Δεν πρόκειται λοιπόν να σας μιλήσω για τις πολύ νέες αυτές ε, μητέρες, στις οποίες αναφερθήκαμε πριν από λίγο. Ομόφωνα όλες αυτές οι γυναίκες είπανε ότι η μετάβαση προς την μητρότητα αποτελεί μια πολύ σημαντική βαθιά αλλαγή, μια αναστρέψιμη για τη ζωή τους. Η ζωή τους δεν άλλαξε εντελώς, αποτελεί μητρότητα μια πολύ μεγάλη πρόκληση, μια πολύ μεγάλη ευθύνη και ορισμένες από αυτές δεν αισθάνονται απαραίτητα έτοιμες για να αντιμετωπίσουν τη μητρότητα. Πάντως όλες μιλάνε για την μητρότητα, για την απόκτηση του παιδιού ως μια πάρα πολύ μεγάλη χαρά που πραγματικά άξιζε τον κόπο. Τους κάναμε την ακόλουθη ερώτηση, αν μπορούσατε να στείλετε ένα μήνυμα προς τον πολιτικό κόσμο προκειμένου να βελτιωθεί η ζωή σας ως μητέρα, ποιο θα ήταν το μήνυμα αυτό. Λάβαμε πάρα πολλές απαντήσεις στο ερώτημα αυτό και βλέπουμε ότι στο σύνολο των απαντήσεων υπάρχει μια κοινή γραμμή. Να τι λένε λοιπόν, τι σας λένε σε εσά, τους βουλευτές, αυτές οι μητέρες. Τρία είναι τα βασικά θέματα τα οποία επαναλαμβάνονται συχνά. Πρώτον, συμφιλίωση της εργασίας με την ιδιωτική ζωή, την οικογενειακή ζωή. Δεύτερον, πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη αναγνώρισης έχουν οι μητέρες αυτές. Αναγνώριση από όλη την κοινωνία, αναγνωριστεί ο ρόλος που διδραματίζουν ως μητέρες. Και τρίτον, μιλάνε για την ανάγκη να έχουν περισσότερο χρόνο για να ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μήνυμα που έχει να κάνει με τη συμφιλίωση επαγγελματική και οικογενειακής ζωής. Οι μητέρες αυτές μιλάνε για τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις ώρες εργασίας και το σχολικό πρόγραμμα, ότι χρειάζονται τις απαραίτητες ποιοτικέ δομές υποδοχής των παιδιών τους. Πολλές φορές μιλάνε για βρεφονιπιακούς σταθμούς στα πλαίσια της επιχείρησης, του χώρου εργασίας. Πολλές ζητάνε κάποιες έμπρακτες οικονομικές λύσεις για να καταφέρουν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στα παιδιά τους. Η συμφιλίωση της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής κατά την άποψή τους δεν θα πρέπει να έχει μόνο ως στόχο την ικανοποιητική ένταξή του στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει παράλληλα να αποτελεί μια αναγνώριση από την κοινωνία για τη σημαντική συμβολή των μητέρων στο λειτουργήμά τους αυτό. Αισθάνονται οι μητέρες αυτές ότι ο ρόλος τους δεν τα γνωρίζετε παρκώ. Θέλουν λοιπόν μια υποστήριξη στο σημαντικότατο αυτό ρόλο που έχουν αναλάβει με τη βοήθεια του πατέρα, προκειμένου να καταφέρουν να συμβάλλουν στην ανατροφή των παιδιών του, προκειμένου να δημιουργήσουν υπεύθυνου πολίτε. Ο ρόλο αυτό προποθέτει μια πολύ συγκεκριμένη υποστήριξη κάθε φορά που οι μητέρε αυτέ είναι μόνε του. Χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να καταφέρουν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση των παιδιών του, ιδίω όταν τα παιδιά αυτά είναι πολύ μικρά το 80% των μητέρων αυτών θα ήθελε να μπορεί να ασχοληθεί πλήρως με την ανατροφή των παιδιών μέχρι να φτάσουν στην ηλικία των τριών ετών, δηλαδή όσον αφορά την προσχολική ηλικία. Όταν τα παιδιά φτάσουν στην ηλικία που μπορούν να πάνε πια στο σχολείο, αλλά ακόμα και στην εφηβεία, θα ήθελαν οι μητέρε αυτέ να μπορούν να επιλέγουν μια ευέλικτη εργασία, να μπορούν να εργαστούν σε ε, καθεστώ μερική απασχόληση. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να είναι πιο κοντά στα παιδιά του κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών. Στην πραγματικότητα δεν καταφέρνουν να υλοποιήσουν τι επιθυμίε του αυτέ και για αυτό το λόγο ζητούν από εσά να λάβετε υπόψη στην ανάγκη του αυτή να ασχοληθούν περισσότερο με την ανατροφή των παιδιών του. Η μεγάλη πλειοψηφία των μητέρων θέλουν να είναι ενεργέ στην αγορά εργασία. Αυτό το οποίο όμω θέλουν παράλληλα είναι σε κάποιε συγκεκριμένε στιγμέ τη ζωή του να μπορούν να έχουν περισσότερο χρόνο για να ασχοληθούν με την οικογένειά του. Θα επανέλθουμε επίσης στην ε, πραγματικότητα που υφίσταται όσον αφορά τους κύκλους ζωής στα πλαίσια μιας οικογένειας. Όσον αφορά το μήνυμα το οποίο θα πρέπει να σταλεί προς τους πολιτικούς, οι γυναίκες αυτές μιλάνε για την κατάσταση που ζουν στα πλαίσια του διαζυγίου, στο ότι θα πρέπει η γονική έρημνα να γίνεται εκ περιπτροπής, στο ότι θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη δικαιοσύνη όσον αφορά την έκθεση στα προβλήματα της δικαιοσύνης, όσον αφορά την φτώχεια, όσον αφορά την πρόσβαση που θα πρέπει να έχουν σε συστήματα υποστήριξης. Οι μόνες αυτές ε, μητέρες διανύουν ένα βίο πολύ πιο δύσκολο σε σχέση με τις μητέρες αυτές που, ζουν, ε, σε που έχουν ένα σύντροφο ή που είναι παντρεμένες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμω να αναγνωριστεί ο ίδιος ρόλος που διαδραματίζουν ως μητέρε, οι ίδιες ανάγκες που έχουν και ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να διαδραματίσουν το ρόλο αυτό τη μητέρα. Πολλές φορές η μείωση, ο μειωμένο χρόνο που έχουν και τα επιπλέον προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν δημιουργούν μεγαλύτερη ένταση, μεγαλύτερε συνθήκε φτώχεια που πολλέ φορέ έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα παιδιά. Τα παιδιά των μόνο γονεακών οικογενειών αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γνωρίζουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των μόνων γονέων ουσιαστικά γυναίκες, μητέρες. Επίσης υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά από την μία μονογονεϊκή οικογένεια στην άλλη. Όλα τα κοινωνικά στρώματα, όλες οι γεωγραφικές περιοχές γνωρίζουν τέτοιες οικογένειες. Το κοινό του σημείο όμω είναι ότι μέσω του χωρισμού και του διαζυγίου πέφτει πολύ σημαντικά το βιωτικό επίπεδο των οικογενειών αυτών. Καλούνται οι μόνοι γονεί να αντιμετωπίσουν ε, τα καθημερινά προβλήματα εντελώ μονομένα, χωρί να υπάρχει υποστήριξη που συνήθω υπάρχει από έναν σύντροφο ή από την οικογένεια. Στην Ευρώπη οι μονογονεϊκέ οικογένειε ε, είναι όλο και περισσότερε. Από το 1968 μέχρι το 2005 το ποσοστό των παιδιών που ζουν με ένα μονογονέα πέρασε από το 6% στο 16%, πράγμα το οποίο αντιστοιχεί σε μία αύξηση του 150%. Η, πλειοψηφία, η πλειονότητα των παιδιών αυτών, το 90% περίπου, ζουν με την μητέρα τους. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε κατε πηγόντω το πρόβλημα αυτό όχι μόνο για τι ίδιε τι μητέρε, αλλά και για τα ίδια τα παιδιά και για το το μέλλον της οικογέν... των κοινωνιών μα. Σα ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που αναλάβατε την πρωτοβουλία σύνταξη ε, μια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρω ότι ε, συντάσσετε εκθέσει και γνωμοδοτήσεις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες οι εκθέσει και νομοδοτήσει αυτέ επηρεάζουν τη ζωή των γυναικών και σα ευχαριστούμε για αυτέ. Καλήσετε την οργάνωσή μου, την ΜΜΜ Ευρώπη, να σα προτείνει κάποιε συγκεκριμένε λύσει. Να, ορισμένε από αυτέ. Πρέπει σαφώ να αυξηθεί ο αριθμός αλλά και η ποιότητα των υπηρεσιών υποδοχής των μικρών παιδιών. Πρέπει όμως παράλληλα να φανταστούμε και νέες λύσεις σε πολλούς τομείς. Θα αναφερθώ σε τέσσερις. Πρώτον, στο χρηματοπιστωτικό τομέα ο φόρος προστιθέμενης αξίας καθώς επίσης και τα οικογενειακά επιδόματα. Θα πρέπει επίσης να αναγνωριστεί μία μη ανιβόμενη εργασία στα πλαίσια της οικογένειας. Σε κοινωνικό επίπεδο τρίτον θα πρέπει να έχουμε μέτρα πρόληψης της διάλυσης της οικογένειας. Θα πρέπει να συμβάλλει περισσότερο σύντροφος ο πατέρας, να βελτιωθούν οι συνθήκες στέγαση των οικογενειών αυτών και να προβλεφθούν μέτρα για τις οικογένειες που μετακινούνται συχνά. Τέλος, θα πρέπει να ενσωματωθούν όλο και περισσότερο οι μητέρες στα τοπικά επίπεδα λήψη πολιτικών αποφάσεων που τις αφορούν περισσότερο. Όσον αφορά το χρηματοοικονομικό επίπεδο, οι ε, μητέρες από τις μονογονιακές οικογένειες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο έκθεση στη φτώχεια θα πρέπει να ζουν σε μια κατάσταση, θα πρέπει να βελτιωθεί το βιωτικό τους επίπεδο. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να αποφύγουμε να μεταφερθεί αυτό ο κίνδυνο φτώχεια και στα παιδιά. Και γι' αυτό το λόγο η οργάνωσή μου συνεργάζεται με άλλε οργανώσεις για την υποστήριξη της οικογένειας και ζητούμε να μειωθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες εκείνες που έχουν να κάνουν με την βρεφονιπιακή ηλικία. Ένα τέτοιο μέτρο τόσο βραχυπρόθεσμο όσο και μακροπρόθεσμο, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρώπη και θεωρώ ότι θα έπρεπε σύντομα να υπάρχει μια ανάλογη σύσταση από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ληφθεί μια τέτοια απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε όλους τους γονείς και κυρίως τους ε, γονείς των μόνο γονεϊκών οικογενειών. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα στέλναμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πολύ χειρό μήνυμα προς όλους τους γονείς εκείνους που μόνοι τους ανατρέφουν τα παιδιά τους, τους μελλοντικούς πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι ορισμένα κράτη-μέλη θα πρέπει να επανεξετάσουν την θεσμική αρχιτεκτονική κοινωνικών υπηρεσιών που έχουν για τα μικρά παιδιά, προκειμένου να, υπάρχει το απαραίτητο πλαίσιο στήριξη του γονέα ήδη από τα πρώτα χρόνια. Χρειαζόμαστε επίση κάποιε καινοτόμε ιδέε για να καταφέρουμε να αναγνωρίσουμε περισσότερα αυτό το οποίο ονομάζουμε child care, την ε, παιδική μέρημνα, την μη αμοιβόμενη αυτή εργασία. Πρόκειται ουσιαστικά για μια εργασία η οποία δεν αξιολογείται χρηματικά, δεν εκτιμάται. Πρέπει λοιπόν να ληφθεί και αυτή η υπόψη στον υπολογισμό του ΑΕΠ μιας χώρας. Αυτή η ανθρώπινη μη αμοιβόμενη εργασία θα πρέπει να αναγνωρίζεται θα πρέπει να εκτιμηθεί προκειμένου να καταφέρει εν τέλει η κοινωνία να συνειδητοποιήσει πόσο σημαντική είναι η συμβολή της και ποιο είναι το ανθρώπινο προσωπικό που αυτή η εργασία απασχολεί. Θέλουμε λοιπόν να εκτιμηθεί, να αποτιμηθεί χρηματικά αυτή η μη αμοιβόμενη εργασία. Η αναγνώριση αυτής της αξίας της μη αμοιβόμενης εργασίας θα οδηγούσε σε κάποιες αποζημιώσεις ή επιδόματα για τις γυναίκες αυτές που ανατρέφουν τα παιδιά τους. Επίσης θα οδηγούσε σε μια μεγαλύτερη συμβολή του συντρόφου, του πατέρα και αυτόν τον τρόπο θα βελτιωνόταν η κατάσταση τόσο για τις μητέρες όσο και για τα παιδιά και ιδιαίτερα για τις μητέρες οι οποίες έχουν χωρίσει ε, και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι εδώ πέρα υπάρχουν διαφορετικοί κύκλοι όσον αφορά την οικογενειακή ζωή. Η περίοδος 25 με 40 έτη είναι η περίοδος εκείνη όπου οι γονείς επομίζονται, όλο και περισσό, περισσότερες ευθύνες για την αντροφή των παιδιών. Επίσης, θα πρέπει να υιοθετήσουμε κάποια μέτρα προκειμένου να μπορούμε να προλαμβάνουμε, αν θέλετε, αυτό το οποίο ονομάζουμε διάλυση τη οικογένεια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την έλλειψη χρόνου, το, τα οικονομικά προβλήματα τα οποία πάρα πολλές φορές προκύπτουν και που δημιουργούν μεγαλύτερη ένταση στα πλαίσια της οικογένειας. Στα πλαίσια της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα και στα κοινωνικά ζητήματα, όχι μόνο στα οικονομικά. Θεωρώ λοιπόν θα πρέπει κάποιες καινοτόμες ιδέες να εγκριθούν για τη στήριξη των οικογενειών σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης πολλές φορές είναι οι οικογένειες αυτές που λειτουργούν ως καταφύγιο προκειμένου να καταφέρουν να διανύσουμε την κρίση αυτή ως το δυνατόν πιο ανώδυνα. Επίσης η οργάνωσή μου πιστεύει ότι θα πρέπει να γίνει και μία έρευνα για τις βέλτιστες εκείνες πρακτικές που υιοθετούνται από ορισμένε χώρες για την υποστήριξη των οικογενειών και για τη μεγαλύτερη συμβολή του πατέρα ήδη από τη γέννηση του παιδιού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις που δεν έχουν γίνει όμως τα περισσότερα κράτη-μέλη, προκειμένου να εξασφαλιστούν αξιοπρεπή χώροι στέγασης, αξιοπρεπής χώροι στέγασης, αξιοπρεπής σπίτια, κατοικίες για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας και την κινητικότητα, της, ε, τη μετατόπιση που μπορεί να οδηγήσει σε μια οικογένεια, ο χωρισμός ή το διαζύγιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, για παράδειγμα, να υπάρχει μια διασυνοριακή αναγνώριση της καταβολής της διατροφής και επίση θα πρέπει να υπάρχει και μια συνεργασία πιο συγκεκριμένη, πιο στενή ανάμεσα στην χώρα προέλευσης και τη χώρα προορισμού του γονέα της μονογονεϊκής οικογένειας. Θα πρέπει η Ευρώπη να προστατεύσει και να υποστηρίξει περισσότερο τις οικογένειες προκειμένου να μην υπάρχουν χωρισμοί, προκειμένου να αποφευχθούν τα διαζύγια για τις δύσκολους καιρούς η οικογένεια αποτελεί το τελικό καταφύγιο. Τέλος, προτείνουμε να σωματωθούν περισσότερο οι μητέρες στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, πολιτικών αποφάσεων. Στην πράξη θέλουμε να γίνει κάτι τέτοιο και σε τοπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, σε κάποιες δύσκολες περιοχές, στα δύσκολα λεγόμενα προάστια των Παρισίων, έχουν δημιουργηθεί κάποια κέντρα, κάποιες αντένες από τη δική μου την οργάνωση, την ΜΜΜ Γαλλίας. Έχουμε λοιπόν εκπροσώπους από την οργάνωσή μου που έρχονται σε άμεση επαφή με τις μητέρες και συστάνε μαζί τους για ζητήματα ανασφάλειες, για ζητήματα εγκληματικότητας, για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Από κοινού προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε λύσεις στα προβλήματα αυτά. Στην καρδιά λοιπόν των κοινοτήτων στις οποίες ζουν, οι μητέρες αυτές μπορούν να φροντίσουν καλύτερα τα παιδιά τους και θέλουν να δημιουργήσουν ένα πιο ασφαλέ περιβάλλον για την ανατροφή του. Κατά αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να σημειώσουμε πρόοδο με τρόπο αποτελεσματικό και συγκεκριμένο και πέρα από οποιαδήποτε ιδεολογία, αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι οι μητέρες ζητούν από εσά να βρείτε καινοτόμε εφάνταστες λύσεις προκειμένου να καταφέρουν να βελτιώσουν την κατάσταση στην οποία ζουν οι ίδιες και τα παιδιά τους και θέλουν μια μεγαλύτερη αναγνώριση και υποστήριξη από την κοινωνία. Κυρία Ματέρα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε τη φωνή των γυναικών εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε Πρόεδρε Κέρκ. Και τώρα η δεύτερη προσκεκλημένη μας, Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Ένωσης Μόνων Γονέων του Βερολίνου στη Γερμανία, Θυμίζω ότι αυτή η Ομοσπονδιακή Ένωση ιδρύθηκε το 1967 ως Ένωση Μόνων Μητέρων. Σήμερα ε, είναι τουλάχιστον 9.000 τα μέλη σε εθνικό επίπεδο και ε, καλύπτει τα συμφέροντα τριών εκατομμυρίων μονογονεϊκών οικογενειών. Δίνω λοιπόν το λόγο στην Πέγγι Λίμπης. Σας συμνιστώ όσο το δυνατόν να μην μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα γιατί δυσκολεύονται διερμηνεί. Εάν θέλετε λοιπόν να τηρήσετε το χρόνο τη ομιλία σα μεν, α φτάσετε και τα 17, αλλά όχι τόσο γρήγορα που να μην μπορούν να σα παρακολουθήσουν οι διερμηνεί. Fast. Yes, I will. <laughs> If it's okay. I prepared... Είχα προετοιμαστεί να μιλήσω αγγλικά Σα ευχαριστώ. Εγώ δεν είμαι η πρόεδρο ή η διευθύντρια αυτής της οργάνωσης που λέγεται Ομοσπονδιακό Σύνδεσμο Μονογονεϊκών Οικογενειών. Είναι μια ΜΚΟ, που υπάρχει από το 1965 και ίδρυσε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο μονογονεϊκών οικογενειών το 2007. Οπότε έχουμε κάποιες έπαφες με ευρωπαϊκές ΜΚΟ που εργάζονται με μονογονικές οικογένειες, ε, επαφές π.χ. με την Ισπανία, Αυστρία, Ελβετία και Σουηδία. Και ε, προσπαθούμε να βρούμε και άλλες οργανώσεις. Η προσέγγιση της οργάνωσής μου, του Ομοσπονδιακού Συνδέσμου Μονογονικών Οικογενειών, είναι να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες στις μόνες μητέρες και πατεράδες και όχι να τους βοηθήσουμε άμεσα. Έχουμε δηλαδή να τους βοηθάμε π.χ. στο να διαχειριστούν ένα μικρό προπολογισμό που οδηγεί στη φτώχεια. Και εδώ πέρα δηλαδή στο βασικό πρόβλημα της γερμανικής πολιτικής που είναι η πολιτική της αγοράς εργασίας. Το να βοηθήσουμε κάποιον στην μεμονωμένη του κατάσταση από την Χάνη, γιατί δεν μπορούμε να μεταφέρουμε αυτά τα ίδια συγκεκριμένα μέτρα σε άλλο άτομο. Όσο δεν υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές που να γίνουν προδιαγραφές και νόμος, δεν θα υπάρχει σημαντική αλλαγή στην όλη κατάσταση. Ποια είναι η κατάσταση λοιπόν των μητέρων που είναι μόνες τους. Στη Γερμανία να είναι κάπως διαφορετικά, αλλά σε γενικές γραμμές έτσι είναι τα πράγματα. Περισσότερε περισσότερες βλέπετε είναι οικογένειες με δύο γονείς, μετά έχουμε 19% μητέρες μόνος τους και 9% ζευγάρια που συγκατοικούν, ε, αλλά είναι ανήπαντρα και έχουν παιδιά. Περισσότεροι γονείς έχουν ένα παιδί, μιλάμε για τα 2 τρίτα περίπου, γύρω στο 70%, ένα άλλο 25% έχουν δύο παιδιά και ένα 6,5% έχουν τρία παιδιά και παραπάνω. Οπότε περισσότερο έχουν ένα ή δύο παιδιά. Και μιλάμε για μητέρες μόνες τους. Οι πατεράδες συνήθως έχουν μεγαλύτερα παιδιά, μεταξύ 10 και 15 ετών ή 15 και 18. Εδώ πέρα βλέπετε το εισόδημα των των μητέρων αυτών, στα δύο τρίτα ε, έχουν λιγότερο από 1500 ευρώ για τον οικοκυριό τους. Και αυτό το διάγραμμα δείχνει πως έχει αυξηθεί η φτώχεια τα τελευταία 10 χρόνια. Βλέπετε στα δεξιά μονογονεϊκές οικογένειες και από την άλλη μεριά ε, παντρεμένες, οπότε βλέπετε τεράστια αύξηση της φτώχειας. Δεν ξέρουμε τι προκαλεί την εξαίρεση, αλλά θα προσπαθήσουμε να τη βρούμε. Οπότε ποια είναι η κατάσταση των μητέρων, των μόνων μητέρων. Όπως όλες τις χώρες της Ευρώπης είναι φτωχές, οι μόνες μητέρες έχουν εισόδημα κάτω του μέσου όρου, οι περισσότερες με ένα ή δύο παιδιά. 40% είναι άνεργες, οι εργαζόμενες φτωχές και ζουν από την πρόνοια. Η υγεία τους είναι χειρότερη από τις παντρεμένες μητέρες και η υγεία των παιδιών τους. Το χάσμα των φύλων στην αμοιβή ε, Στη Γερμανία είναι 23%, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα στοιχεία του 2008 λένε ένα 13%. 29,3% των εργαζόμενων γυναικών είναι στον χαμηλόμισθο τομέα, δηλαδή στις υπηρεσίες. Πολιτικές και λύσεις. Για να βελτιωθεί η κατάσταση για τις ανήπαντρες μητέρες πρέπει να αναλυθούν οι αιτίε. Υπάρχουν πολλές αιτίε που έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία χρόνια. Ο βασικός λόγος είναι ανεργία σε part part-time, χαμηλή μισθή, υψηλή φόρη, δεν υπάρχει φροντίδα για τα παιδιά και βεβαίως δεν υπάρχει και διατροφή από πλευράς του άλλου γονέα. Η γερμανική κυβέρνηση επικεντρώνεται σε δύο πολιτικές άμεσες πληρωμές, δηλαδή επίδομα παιδιού και προγράμματα για να ενταχθούν οι άνθρωποι στην αγορά εργασίας. Το Εθνικό Υπουργείο Εργασία έχει ξεκινήσει αρκετά προγράμματα για να ενταχθούν κάποιε ομάδε του πληθυσμού στην αγορά εργασία, π.χ. για μετανάστε, για ανάπηρου και για μακροχρόνια ανέργου. Υπάρχει εστίαση στις μονογονεϊκές οικογένειες επειδή πολύ μεγάλη ομάδα, γύρω στα 630.000 άτομα, δεν έχουν βρει δουλειέ που να πληρώνουν επαρκώ εδώ και χρόνια παρά τι δραστηριότητε του ΑΕΔ ένα τριετές πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που λέγεται «Καλές δουλειές για μονογονεϊκές οικογένειες». Έχει ξεκινήσει ειδικά για τους γονείς εκείνους που έχουν μόνιμη ενεργεία και 95% είναι μητέρες και ζουν από τα τις κοινωνικές παροχές. 60 ε, εκατομμύρια ευρώ θα πάνε σε 79 όργα, έργα με σε ολόκληρη τη χώρα για να ενταχθούν περισσότερες μητέρες στην αγορά εργασίας με στόχο να αυξηθούν οι πιθανότητε των μόνων γονιών να βρουν δουλειές με το να βελτιωθούν τα κέντρα εργασίας ε, του ΑΕΔ, να αυξηθούν τα προσόντα των γυναικών αυτών και οι υπηρεσίε φροντίδα των παιδιών. Θα ήθελα τώρα να πω κάτι για τι άμεσε πληρωμέ και για τα προγράμματα τη αγορά εργασία. Άμεσε πληρωμέ. Ο ΩΣΑ ασκεί συχνά κριτική στην γερμανική πολιτική που είναι η αύξηση του παιδικού επιδόματος, του επιδόματος παιδιών γιατί δεν μειώνει τη φτώχεια. Η UNICEF με την έκθεση Innocenti καταλήγει στα ίδια συμπεράσματα. Μια τρέχουσα γερμανική μελέτη από το Ίδρυμα Hans Beckler δείχνει συγκεκριμένα πως τα τρέχοντα μέσα οικογενειακής πολιτικής αποτυγχάνουν στην προσπάθειά τους να μειώσουν τη φτώχεια. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι πως υπάρχουν πολλά διαφορετικά προγράμματα. Υπάρχει αυξανόμενο κίνημα ΜΚΟ στη Γερμανία που προτείνουν να αλλάξει θεμελιωδώς το σύστημα στήριξης των οικογενειών τα έργα τώρα στην αγορά εργασίας. Υπήρχαν διάφορα έργα για τις ανήπαντρες μητέρες τα τελευταία 20 χρόνια, τα οποία έχουν αναλυθεί σε μία μελέτη των Κουλ και Ρίτ Κατέληξαν στο συμπέρασμα και η οργάνωσή μου πιστεύει, μαζί με πολλές άλλες, πως έχουν δίκιο, πως δεν θα υπάρχει καμία επιτυχία συμμετοχής των ε, μόνων γυναικών στην αγορά εργασίας όσο υπάρχει τόσο μεγάλη ανισότητα, κάτι το οποίο σημαίνει πως οι ανήπαντρε μητέρε έχουν λιγότερες πιθανότητε να βρουν δουλειά. Όχι επειδή είναι ανήπαντρε μητέρες, αλλά πρώτα απ' όλα είναι γυναίκες και δεύτερον επειδή είναι μητέρες. Βασική προσπάθεια δεν θα πρέπει να είναι να κάνουμε το ένα πρόγραμμα μετά το άλλο και να παρουσιάζουμε έτσι διάφορα ωραία σοου και βέλτιστες πρακτικέ παρά το ότι αυτό δεν έχει πραγματικά αποτελέσματα μετρήσιμα. Τα περισσότερα από τα μέτρα αυτή τη στιγμή είναι είτε ε, εν εξελίξει στη φάση των βέλτιστων πρακτικών είτε στην αξιολόγηση. Και οι πρώτες εκθέσεις δείχνουν πως κάποια ίσως είχαν θετικά αποτελέσματα σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των αρχών. Και άρα ερχόμαστε στο ερώτημα ποια πρακτική λύση και ποια πολιτική θα έχει αποτελέσματα για να βελτιώσει ουσιαστικά την κατάσταση των ανήπαντων μητέρων. Αυτέ τι μέρε στη Γερμανία έχουμε για πρώτη φορά τα αποτελέσματα μια εμπειρογνωμοσύνη τη πρώτη κρατική έκθεση για την ισότητα ανδρών και γυναικών που είναι στι εφημερίδε. Το βασικό συμπέρασμα είναι πω η πολιτική της γερμανικής κυβέρνησης αποτρέπει τις γυναίκες από το να εκμεταλλευτούν πλήρως το δυναμικό τους και βασικό είναι να καταρριφθούν λεγόμενες μήνυ δουλειές και να μεταρρυθμιστεί το φορολογικό σύστημα. Δηλαδή να υπάρξει ελάχιστος βασικός μισθός, να υπάρξει ποσόστοση για γυναίκες και στις ε, ηγετικές θέσεις, να σκεφτούμε πώς θα μπορέσουμε ο χρόνος εργασίας να φιλικό στην οικογένεια και βεβαίως ε, να βελτιωθεί το σύστημα της διατροφής των παιδιών. Υπάρχουν και πάρα πολλέ άλλε στάσεις που κατά βάση, κατά την άποψή μα αφορούν την ισότητα. Η ισότητα είναι αυτό το οποίο λείπει από τη Γερμανία, από πλευρά εκπαίδευση υγεία, φροντίδα των παιδιών, καριέρας και φίλου κοινωνικού. Οπότε χαιρόμαστε για το ότι μόλις δημοσιεύτηκε από την πλατφόρμα την οικογενειακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα ερευνητικό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια έκθεση η οποία αναφέρει την ισότητα ως μία από τις βασικές διαστάσεις της ε, ποιότητας οικογένειας. Και αναφέρω κατά λέξη. Η ισότητα είναι βασικό στόχος της σύγχρονης ε, ευρωπαϊκής ε, κοινωνίας και διατρέχει όλα τα άλλα ζητήματα. Γίνεται αντιληπτή με την πολύ γενική έννοια, δηλαδή όλα τα άτομα να έχουν τι ίδιε ευκαιρίε να συμμετέχουν στην κοινωνία με κάθε δυνατό τρόπο και σε κάθε επίπεδο. Το συμπέρασμά μου. Οι οργανώσει μονογονεϊκών οικογενειών δεν βλέπουν να υπάρχει ε, αηφορία στην επίτευξη αποτελεσμάτων από τα έργα αυτά. Το να επιλέγουμε μητέρες όπως η με συγχωρείτε, όπως οι ανήπαντρες μητέρες ε, για τις πολιτικές μας μας βοηθάει να αντιληφθούμε γιατί αποτυγχάνουν οι πολιτικές και γιατί έχουμε τα προβλήματα, αλλά δεν αλλάζει τις δομές που προκαλούν την ανισότητα. Υπάρχουν πάρα πολύ καλές ιδέες που προκύπτουν από την έρευνα και τα πολιτικά μέσα για να εγγυηθούμε την συμμετοχή και βεβαίως ε, να ε, απελευθερώσουμε τα άτομα όταν έχουν κάποιε ευθύνε. Οπότε εμεί θεωρούμε πω η πολιτική πρέπει να ξεκινήσει σήμερα. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, Λίμπης. Και τώρα για να έχουμε και την συνεισφορά της, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε την κυρία Παρασκευά και πάλι. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. θα Ήθελα να είμαι σύντομη, αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα να εστιαστώ σε κάτι το οποίο είπαν οι κυρίες Δελίδε Κέρκη και Λίμπιχ. Πρώτα απ' όλα να αναφερθώ στο ζήτημα της φτώχειας της παιδικής. Όπως ανέφερα πριν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη θέση πως όλα τα παιδιά πρέπει να ωφεληθούν από επιδόματα καθολικά και συγκεκριμένους στόχους μετά ανάλογα με το ποιος τα χρειάζεται περισσότερο λόγω της κατάστασής του. Και στο πλαίσιο αυτό θεωρώ πως τα παιδιά τα οποία ζουν σε οικογένειες μόνο γονοϊκές και αυτά που ζουν σε οικογένειες με πάνω από τρία παιδιά αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κίνδυνο να ζουν σε φτώχεια. Και άρα θα πρέπει να είναι ένας από αυτούς τους στόχους. Το ζήτημα της απλήρωτης εργασίας. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο εδώ και πολλά χρόνια μας απασχολεί στη μονάδα ισότητας των φύλων, ειδικά ε, όσων φροντίζουν κάποια άλλα μέλη της οικογένειας και δεν μιλά μόνο για παιδιά, αλλά και τους ηλικιωμένους και άλλα εξαρτώμενα μέλη. Και νομίζω πως είναι ένα ζήτημα στο οποίο θα επανέλθει η Κομισιόν. Ένα τρίτο ζήτημα που δεν ανέφερα, αλλά προέκυψε την προηγούμενη εβδομάδα στην Επιτροπή σας με την υιοθέτηση της έκθεσης του γυναικείου προσώπου της φτώχεια είναι το ζήτημα του ελάχιστου εισόδηματο. Και εκεί πέρα θεωρώ πως η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει δράση έτσι ώστε να υπάρξει ένα ελάχιστο εισόδημα για όλους για όλες. Αυτή τη στιγμή όλες οι χώρες πλην Ελλάδας, Ιταλίας και Ουγγαρίας έχουν ένα τέτοιο ελάχιστο εισόδημα όμως περισσότερες χώρες είναι τόσο χαμηλό που δεν επιτρέπει να ξεφύγουν οι άνθρωποι από τη φτώχεια. Χρειάζεται λοιπόν ένα ελάχιστο εισόδημα, το οποίο θα επιτρέψει στους ανθρώπους να ζουν με αξιοπρέπεια. Επίσης, όπως αναφέρθηκε, τα μετρητά δεν είναι πανάκια στο πρόβλημα. Όλο αυτό το πρόβλημα του συμβιβασμού θα πρέπει να το ξαναδούμε για να επιτρέψουμε να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένες ανάγκες των μόνον γονέων. Υπάρχουν πολλά καλά παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών. Θα ήθελα να αναφέρω παραδείγματος χάρη το πρόγραμμα Τζεπέτο που ξεκίνησε πρώτα απ' όλα στη Φιλανδία και μετά στη Γαλλία και αλλού όπου υπάρχουν 24 ε, ώροι παιδική σταθμή όπου οι γονείς ε, μπορούν να βρουν στήριξη. Θα ήθελα επίσης να τονίσω τη σημασία της αναγνώρισης του ρόλου των οικογενειών στην ανατροφή των παιδιών. Και εγώ είμαι γονιός και συχνά τίνουμε να λέμε πως το σχολείο πρέπει να κάνει αυτό, το σχολείο πρέπει να κάνει το άλλο. Όχι. Είμαστε γονείς και πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Και τέλος αλλά εξίσου σημαντικό θα ήθελα να ανακοινώσω πως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας κατά της στόχιας σκοπεύουμε να έχουμε μια σύσταση για το πώς θα προληφθεί και θα αντιμετωπιστεί η παιδική φτώχεια που θα αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ζητήματα και η σύσταση αυτή προβλέπεται να υιοθετηθεί το 2012. Νομίζω λοιπόν πως αυτά είναι τα βασικά ζητήματα επί των οποίων θα μπορούσε να απαντήσει η Κομισιόν. Και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και πάλι το Κοινοβούλιο για την πρωτοβουλία που ανέλαβε και ελπίζουμε να συνεχίσει παραπέρα. Ευχαριστώ. Οπωσδήποτε θα το πράξουμε. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα να δώσουμε το λόγο στις συναδέλφους για παρεμβάσεις και ερωτήσεις προς τις εμπειρογνώμονες. Δίνω το λόγο στην κυρία Ήλντα Φιγκέιρα εδώ, εισηγήτρια εκ μέρους της ε, ομάδας της ΒΟΕ. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε. Με συγχωρείτε που καθυστέρησα κάπως, αλλά υπήρχε ένα θεματάκι με την πτήση που έφτασε καθυστερημένη κι αυτή. Θεωρώ ότι το θέμα αυτό είναι σημαντικό. Διότι στο πλαίσιο των διακρίσεων κατά των γυναικών, το ζήτημα των γυναικών που μόνες μεγαλώνουν τα παιδιά τους λαμβάνει διαστάσεις ανησυχητικές. Οι εργαζόμενες ή οι άνεργες όταν έχουν και τα παιδιά τους να αναθρέψουν και είναι και μικρά το θέμα είναι τεράστιο. Ξέρω πάρα πολλέ περιπτώσει όπου αυτέ οι περιπτώσει μετατρέπονται σε πραγματικέ τραγωδίε. Όμω, στην ε, παρούσα φάση, όπου σε ορισμένε χώρε, όπω για παράδειγμα στην Πορτογαλία, αυτή την κατάσταση γνωρίζω καλά γιατί από εκεί προέρχομαι, αλλά και αλλού, όπως στην Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία και σε πολλές άλλες χώρες, η φτώχεια αυξάνεται δραματικά. Περικοπές στην κοινωνική πρόνοια είναι αναπόφευκτες. Το ίδιο και τα, τα επιδόματα τα οικογενειακά. Συμπεριλαμβανομένων των, στηρι... συμπεριλαμβανομένων των στηρίξεων προς τις μονογονεϊκές οικογένειες και τις γυναίκες που ζουν με τα παιδιά τους μόνες, με χαμηλούς μισθούς, με προσωρινή εργασία. Οι καταστάσεις αυτές είναι δραματικές. Την περασμένη μόλις εβδομάδα είδαμε εδώ να οργανώνεται στην αγορά μια συζήτηση για την φτώχεια και διά, διάφοροι οργανισμοί ζήτησαν από εμάς τους βουλευτές να μεταφέρουμε στους συναδέλφους μας την οργή για τα όσα συμβαίνουν στο κοινωνικό τομέα. Την επιδείνωση της φτώχειας, την επιδείνωση, την όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Φτώχεια που φτάνει πλέον πολύ συγκεκριμένε κοινωνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, αλλά και τα παιδιά, τους νέους, τα ποσοστά ανεργίας σε ορισμένες χώρες ξεπερνούν το 45%. Η δραματική κατάσταση λοιπόν αυτή αξίζει όλη μας την προσοχή. Ε, αυτό που θέλω εδώ είναι πραγματικά να κάνω αυτό που τους υποσχέθηκαν, να μεταφέρω την μεγάλη αυτή ε, δυσαρέσκεια, την οργή των πολιτών για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που αυξάνεται η φτώχεια και που θίγει πλέον και τομεί όπως αυτός που σήμερα συζητούμε. Την ομάδα δηλαδή των γυναικών που ζουν μόνες. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε όμως και για τις ηλικιωμένε γυναίκες. Είναι η πλειοψηφία μεταξύ των ηλικιωμένων. Και οι περισσότερες έχουν συντάξεις πολύ χαμηλές εξαιτία της χαμηλής μισθοδοσίας εξ αρχής, Εξαιτία των προσωρινών θέσεων εργασία, τη μητρότητα. Μιλάμε για γυναίκες με πολύ χαμηλού μισθού που διωγγώνουν τα ποσοστά φτώχειας. Όταν θα φύγουμε από το Ευρωπαϊκό κατά Καταπολέμησης της Φτώχειας και θα δούμε οι δείκτες αυτοί να έχουν αυξηθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα πρέπει να κοιτάμε μόνο τους μέσους όρους. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος συγκερά... μπορεί να συγκεράσει την κατάσταση χωρών που είναι πλούσιες, άλλες που βρίσκονται σε οικονομική ανάπτυξη και άλλες όχι. Και καλύπτει το φρικτό αυτό δράμα κάποιων χωρών που ζουν σε τόσο δύσκολες συνθήκες. Ήθελα λοιπόν οπωσδήποτε να μιλήσω για την όξυνση των ανισοτήτων και την επιδείνωση της φτώχειας. Τα οικονομικά μέτρα που αυτή τη στιγμή σχεδιάζονται, συγκεκριμένα το πακέτο της οικονομικής διακυβέρνησης, νομίζω θα επιτείνει την κατάσταση αυτή. Διότι το να μην λαμβάνουμε υπόψη τις αρχές της αλληλεγγύης, της οικονομικής και κοινωνικής συνεχής, της φτώχειας και όλων αυτών των ζητημάτων, της ανεργίας, όλα αυτά το πακέτο δεν τα πέραν και απουσιάζει από κάθε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, η έννοια αυτή, η συνοχή. Είναι λοιπόν μεγάλη μας ανησυχία αυτό το θέμα. Γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ και συζητούμε και θέλουμε να αφήσουμε κάποιες από αυτές τις εκφράσεις ανησυχίας, επαγρύπνησης, οργής που ακούσαμε και που μας μετέφεραν και κοινωνικές οργανώσεις που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία του Ευρωκοινοβουλίου την περασμένη εβδομάδα. Καλό θα ήταν να τοποθετηθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με ορισμένα από αυτά τα ζητήματα, όμως φτάνει πια και με τα λόγια. Όλοι μας λένε ότι δεν θέλουν πια λόγια, θέλουν πράξεις, ενέργειες, δράσεις. Δεν μπορώ να συνεχίσω κι εγώ να μιλάω λοιπόν. Ας λέμε κάτι αλλά μετά να περνάμε στην πράξη ε, κατώτατος ε, μισθός, πρόταση και δράση. Αυτό ήταν μια σημαντική πρόταση για να καταπολεμήσουμε λόγω χάρη τη φτώχεια φέτος. Την φτώχεια των γυναικών, τη φτώχεια των παιδιών. Είναι ζητήματα συγκεκριμένα, χειροπιαστά. Αυτά θέλω να σκεφτούμε. Ευχαριστούμε κυρία Φεγκουρέιδο. Σα θυμίζω ότι το λόγο έχετε για πέντε λεπτά και το λόγο έχει ακριβώ κυρία Λούλινγκ εκ μέρου του ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ έχω συγκεκριμένε ερωτήσει προ τι εισηγήτριε. Για την πρώτη μα προσκεκλημένη, την πρόεδρο του Διεθνούς Κινήματος Μητέρων, Μα είπε για φάνταστε λύσει πρέπει να εξεύρουμε και μα μίλησε και για ΦΠΑ. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξή. Πώ αντιλαμβάνεστε αυτή τη λύση, Πώ θα είμαστε εφάνταστε στο επίπεδο του ΦΠΑ, Υπάρχουν κανόνε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε ελάχιστα επίπεδα και ελάχιστα επιτόκια. Η μειωμένη επιτόκια. Τα κράτη-μέλη μερικά μπορούν να τα εφαρμόσουν, μερικά όχι. Στην Αγγλία Θυμάμαι την εξαίρεση από, τη ΦΠΑ, από το ΦΠΑ για τα παιδικά υποδήματα και κάτι ανάλογα προϊόντα. Πώς σας αντιλαμβάνεστε αυτή τη λύση σας λοιπόν που να ανακεφάνταστε στο επίπεδο του ΦΠΑ. Επίσης μιλήσατε για τους υπολογισμούς του ΑΕΠ και ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι εργασίε χωρί αμοιβή των γυναικών. Ε, πώς θέλετε να τα μετρήσουμε αυτά ποσοτικά. Εφόσον δεν υπάρχουν αμοιβέ, διότι σίγουρα αυτό θα προκύψει και που το ποσοστό απασχόληση των γυναικών είναι χαμηλότερο. Και έτσι διωγγώνεται το, το ΑΕΠ, ξέρετε ότι υπάρχουν πολλές παροχές και πολλές κυρίως ε, πληρωμές των κρατών μελών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν πόροι που αποδίδονται Οι συνεισφορές δηλαδή των κρατών μελών προς τον ευρωπαϊκό προπολογισμό βασίζονται στο ΑΕΠ. Ε, τώρα δεν είστε να διεκδικήσουμε και να επιβάλλουμε και ποινές στα κράτη-μέλη όπου δεν είναι τόσο ε, διαδεδομένη η άτυπη εργασία. Τώρα για, την, για, τα οικογενειακά επιδόματα. Μα υπάρχουν χώρες όπου αυτό προβλέπεται και είναι και κανονικότατο στην λειτουργία του φαινόμενο, δηλαδή μηνιαίως καταβάλλεται το επίδομα στη μητέρα. Επίσης, μιλήσατε για την οργάνωση των υπηρεσιών ε, φροντίδας των παιδιών, νηπιαγωγείων κλπ. Δεν μπορώ να μην το σχολιάσω αυτό, γιατί το δεκαετία του 80 είχαμε κάνει μια έκθεση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την διοργάνωση αυτών των υπηρεσιών. Νομίζω ότι ισχύουν τα τότε. Δεν χρειάζεται να ξανακάνουμε τα ίδια. Οι συστάσεις μας τότε είχαν εφαρμοστεί. Είμαστε πολύ καλύτερα εξοπλισμένοι τώρα από ό,τι στο παρελθόν. Μιλήσατε και για μια υποδομή 24 ώρες λειτουργίας, για αυτές ακριβώς τις ε, υπηρεσίες, τους σταθμούς φροντίδας των παιδιών. Εγώ σας ρωτώ πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτό αφού λέτε ότι είναι τόσο αναγκαίο. Και για το ρόλο των μητέρων. Ζητήσατε περισσότερο χρόνο για τις μητέρες να λαμβάνετε υπόψη ο κύκλο ζωή επίση. Αλλά και περισσότερη δουλειά ζητήσατε. Εδώ νομίζω ότι μα ζητάτε να τετραγωνίσουμε κάπως τον κύκλο, έτσι. Πώ θα γίνουν όλα αυτά. Πώ θέλετε όλα αυτά να χρηματοδοτηθούν. Πώ θα υλοποιηθούν. Και σε ό,τι αφορά τι στατιστικέ περιφτώχεια. Εδώ προσέξτε λιγάκι. Διότι τις στατιστικές αυτές πρέπει κανείς να τις διαβάζει με μεγάλη επιφύλαξη. Οι στατιστικές για τη φτώχεια στα διάφορα κατημέλη πρέπει να σας πω ότι για το Λουξεμβούργο, λόγω χάρη από που εγώ προέρχομαι εννοείται διαφορετικά. Δηλαδή, ο φτωχό στο Λουξεμβούργο, αν περάσει τα σύνορα, ε, είναι πολύ πλούσιο στη Λορένη. Να προσέχουμε λοιπόν λίγο με τις στατιστικές. Έχουμε αυξημένου αριθμούς βέβαια, έχουμε όμως και κατώτατου μισθού που είναι και πιο αυξημένοι από τις άλλες χώρες. Μιλάμε για 1.800 ευρώ το μήνα, ενώ στη Γερμανία είναι η μόνη επιλογή που έχετε αυτό ο κατώτατο μισθό και αν δεν θέλετε δεν έχετε και καθόλου. Μιλάμε για 800 ευρώ κάποιε φορές και για χώρες που ζητούν εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, τι λέμε τώρα εδώ. Δεν μπορεί να είναι ίδιο το επίδομα αυτό σε όλα τα κάτι μέλη. Οι καταστάσει διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, έτσι. Να ξέρουμε Μήπω μήπως αυτά που διεκδικούμε είναι απατηλά, τελείω τοπικά. Και δεν ξέρω και σε τι διευκολύνουν ακριβώ τι γυναίκε. Έχω και άλλη ερώτηση. Προ την Γερμανίδα εμπειρογνώμονα, γιατί ξέρω ότι στη Γερμανία γίνεται αυτή τη στιγμή μεγάλη συζήτηση για τα θέματα αυτά. Τι πρέπει να γίνει, να προβλεφθούν επιδόματα, πρέπει να δίνουμε χρήμα ή να προσφέρουμε υπηρεσίες. Νομίζω ο καθένας θα πρέπει να είναι υπεύθυνο των επιλογών του. Όμως είναι σαφές ότι τα κονδύλια που φτάνουν, τα χρήματα που φτάνουν στα έστω μέσω υπηρεσιών, αλλά στα παιδιά, είναι κάτι που ήδη το έχουμε προβλέψει με ψηλότατα επιδόματα, με υπηρεσίες που περνάχαν από επιταγές στα, στις ενδιαφερόμενες Εδώ υπάρχει όμως και η αρχή της επικουρικότητας. Δεν μπορούμε να πάρουμε ένα ενιαίο μέγεθος για όλους, one size fits all για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Τόμψον και θα παρακαλέσω τις συναδέλφους να σεβαστούν το χρόνο. Ε, Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σχολιάσω αυτό το οποίο είπε η κυρία Λίμπης. Γιατί νομίζω πως ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο ακούστηκε ότι το θέμα αφορά το φύλλο το να είναι κανείς γυναίκα και μητέρα. Και άρα οι μητέρες, οι ανήπαντρος είναι σε κακή θέση στη Γερμανία. Αυτό είναι σωστή προσέγγιση. Γιατί βλέπετε πως γενικώ οι γυναίκες στη Γερμανία έχουν από τις χειρότερες συνθήκες στην αγορά εργασίας. Δουλεύουν part-time, πληρώνονται χαμηλά, δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί Δηλαδή το να εργάζεται κανείς στη Γερμανία ε, δεν είναι το ίδιο παντού. Είναι άλλο να δουλεύει κανείς στη Volkswagen και άλλο να είναι γυναίκα στις υπηρεσίες. Οπότε συμφωνώ μαζί σας σε αυτό, αλλά δεν νομίζω πως ε, ο βασικός μισθός, ο ελάχιστος μισθός είναι η λύση σε κάποιες χώρες στην Ευρώπη. Εμείς υποστηρίζουμε το ελάχιστο εισόδημα στο δανέζικο κόμμα, αλλά όχι τον ελάχιστο μισθό. Ε, το ελάχιστο εισόδημα πρέπει να βασίζεται στο ΑΕΠ των διαφόρων χωρών. Ο ελάχιστος μισθός είναι θέμα της αγοράς εργασίας. Αλλά ήδη στη Γερμανία έχει ελάχιστο εισόδημα με το σύστημα Hartz 4, οπότε κάποια λεφτά έχετε το μήνα. Ε, βεβαίως αυτό θα επηρεάσει τους ε, του γονείς. Όσον αφορά την οικογενειακή πολιτική φοβάμαι πως θα υπάρχει λιγότερη οικογένεια στο μέλλον. Γιατί λόγω και των δημογραφικών τάσεων. Όπως μελετάμε την αγορά εργασίας μπορούμε να δούμε και την αγορά του γάμου ας πούμε. Γιατί η κατάσταση όπως έχει σήμερα και γίνεται όλο και περισσότερο έτσι, στις μεγάλες πόλεις βλέπουμε περισσότερες γυναίκες από άντρες και στις απομακρυσμένες περιοχές βλέπουν περισσότερους άντρες από γυναίκες. 70% σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες είναι οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων, οι γυναίκες. Δεν θέλουν να παντρευτούν έναν μαραγκό, αλλά δεν μπορούν να παντρευτούν και απόφυτο πανεπιστημίο, οπότε τι κάνουν, ζουν μόνες τους και υιοθετούν ή κάνουν τεχνητή γονιμοποίηση. Και στη χώρα μου αυτό είναι διάκριση. Έχουν κάνει νομοθεσία και είναι ενδιαφέρον αυτό να το δει η Κομισιόν, όπου λένε κάθε ανήπαντρη μητέρα έχει δικαίωμα σε κάποιο καθολικό επίδομα, αλλά εάν έχει κάνει τεχνητή γονιμοποίηση ή έχει οθετήσει, ή διαλέγεις να είσαι ανήπαντρη μητέρα, τότε δεν επιτρέπεται να έχεις το διπλό αυτό επίδομα όπως οι άλλες ανήπαντρες μητέρες. Αυτή είναι νέα τάση και βλέπουμε πώς αγιαλεύουν διαλέγουν οι γυναίκες να ζουν στο μέλλον. Ε, και αυτό το οποίο είπαμε πριν για την Ιταλία, ότι αντί για το κράτος φροντίζει η οικογένεια. Εγώ συνάντησα όταν ήμουν νέα μια γυναίκα από τη Χιλή στη Δανία. Ήταν πρόσφυγας και είχε ενοποίησε την οικογένειά της, δηλαδή ήρθε και ο άντρας της εκεί πέρα και όταν ήρθε ο σύζυγος είχε παντρευτεί μια άλλη. Και τη ρώτησα, μα γιατί δεν επιστρέφεις στη Χιλή, από όπου μας ήρθες κιόλα στην οικογένειά σου. Και μου είπανε, τότε θα ανήκα πάλι στον πατέρα μου. Χωρίς άντρα δεν είσαι τίποτα. Και σε ελέγχει ο πατέρα σου, ο αδερφός σου, Νομίζω τουλάχιστον οι γυναίκες στην Ευρώπη πρέπει να έχουν την επιλογή για το τι θα κάνουν. Ε, πρέπει να είναι δηλαδή βασικό δικαίωμα να έχουν μια συνεισφορά από τον πρώην σύζυγο και να αποφασίζουν μόνες τους τι θα τα κάνουν. Ευχαριστούμε την κυρία Τόμψον και τώρα εμπειρογνώμονές μας για το συμπέρασμα. Και να σας πω και μια καλή είδηση. Έχετε περισσότερα από 10 λεπτά σχεδόν. Πρώτα απ' όλα η κυρία Λίντα η πρόεδρος του κινήματος των μητέρων. Να απαντήσω πρώτα στην κυρία Λούλινγκ. Αυτό το οποίο έκανα είναι ότι σας μετέφερω σαστικά τα όσα που μας έχουν πει οι μητέρες μέσω των ερευνών, μέσω των ατελιέ, των εργαστηρίων που έχουμε οργανώσει ζήτησαν περισσότερο χρόνο, ζήτησαν μεγαλύτερη αναγνώριση των δυσκολιών που έχουν στο να συνδυάσουν επαγγελματική και οικογενειακή ζωή με βάση τον οικογενειακό κύκλο ζωής στον οποίο βρίσκονται. Σαφώς θέλουν να εργαστούν, θέλουν να εργάζονται περισσότερο όταν έχουν μεγαλώσει όμως τα παιδιά τους, λιγότερο όταν τα παιδιά είναι μικρότερα. Εγώ απλώς αυτό που έκανα είναι ότι σας μετέφερα τα όσα μας έχουν πει οι μητέρες αυτές μιλάνε όλο και περισσότερο για το ρόλο που έχουν ως μητέρες, με ιδιαίτερη ανησυχία, γιατί για αυτές αποτελεί σημαντικότατη προτε... προτεραιότητα. Αυτό δεν σημαίνει δεν θέλουν να εργαστούν. Επιθυμούν κάποια στιγμή να αναγνωριστεί όμως το γεγονός ότι υπάρχουν στιγμές στη ζωή τους που η οικογένεια είναι πιο σημαντική και άλλες στιγμές που είναι σε θέση να εργαστούν περισσότερο. Αυτή είναι η βασική επιθυμία την οποία εκφράζουν. Γιατί ξέρετε ότι στην πραγματικότητα οι μητέρες δεν μπορούν να κάνουν ακριβώς αυτό το επιθυμούν να κάνουν γιατί δεν είναι έτσι η ζωή. Τώρα, για τις εφάνταστες αυτές λύσεις, φόρος προστιθέμενης αξίας. Πρόκειται για ένα αίτημα το οποίο ακούσαμε πάρα πολλές φορές τα μηνύματα τα οποία στέλνουμε προς πολιτικούς. Ορισμένοι πιστεύουν ότι από τη στιγμή που ανατρέφουμε εμεί τα παιδιά και τους πολίτες του αύριο θα πρέπει να έχουμε και μία βοήθεια για αυτό το πράγμα. Αυτά είναι τα βασικά σχόλια τα οποία έχουμε ακούσει. Σίγουρα δεν είμαι εμπειρογνώμων, δεν ξέρουμε ακριβώ με ποιο μηχανισμό θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κάτι τέτοιο. Πάντω, το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσαν να κάνουν μια κάποια σύσταση στα κράτη-μέλη, την οποία στη συνέχεια αυτά μπορούν να ακολουθήσουν ή όχι. Το βασικό πάντω μήνυμα είναι ότι θα καταφέρουμε να πούμε προ τι οικογένειε ότι κοιτάξτε, το ότι ανατρέφεται παιδιά είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα παιδιά αυτά θα είναι μελλοντικοί πολίτε τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντοποιούμε ότι καταβάλλεται προσπάθειε για την ανατροφή του και συντοποιούμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε. Σίγουρα εμεί δεν μπορούμε να σα δώσουμε έμπρακτα μία απάντηση, δεν μπορούμε να σα πούμε ακριβώ πώ θα μπορούσαν τα πράγματα να διοργανωθούν. Κάνουμε απλώ μία σύσταση. Τώρα, μία αμοιβόμενη εργασία. Έγινε ήδη μία έρευνα για την μία αμοιβόμενη αυτή εργασία, αλλά με τρόπο κατακαιρματισμένο σε διάφορες χώρες. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ποσοτικοποιήσουμε τα πορίσματα των ερευνών αυτών, προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα το οποίο θα υπογραμμίζει την σημασία της μία αμοιβόμενης αυτής εργασίας, για να γνωρίσουμε την αξία της εργασίας αυτής. Αν διαβάσετε τα πορίσματα της έρευνας, θα δείτε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι μητέρες οι οποίες έχουν απαντήσει σε ερωτηματολόγια μας λένε ότι δεν αναγνωρίζεται από την κοινωνία ο ρόλος μας. Μόνο και μόνο το να καταφέρουμε να αναγνωρίσουμε και να αποτιμήσουμε από οικονομικής πλευράς τη μία αμοιβόμενη αυτή θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αν καταφέρουμε μάλιστα να την αναγνωρίσουμε επίσημα και οικονομικής πλευράς, τότε σαφώς θα μπορούν να υπάρξουν και μέτρα από τους πολιτικούς τόσο για τις μητέρες όσο και για τους πατέρες. Δεν μίλησα για τα οικογενειακά επιδόματα προς τις μητέρες, δεν μίλησα για την δομή αυτή υποστήριξης 24, 24 ώρες το 24ωρο. Σε σχέση αυτά που είπε η κυρία Τόμσον, μπορώ να πω ότι οι οικογένειες, τουλάχιστον οι μητέρες, θέλουν να μπορούν να ασχοληθούν περισσότερο με την οικογένειά τους, αλλά στα πλαίσια ομαλών συνθηκών, όχι στα πλαίσια δυσκολιών και προβλημάτων. Αυτό το οποίο ζητάνε είναι να μπορούν να ασχοληθούν περισσότερο και πιο ποιοτικά με τις οικογένειές τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα για τα συμπεράσματά της να δώσουμε το λόγο στην πρόεδρο Λίμπης. Θα μιλήσω γερμανικά. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε τρία ζητήματα. Πρώτα απ' όλα να αναφερθώ σε αυτό το οποίο ακούστηκε για τη μεγάλη κοινωνία και την κυρία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ανέφερε τη σκέψη για μια βασική ασφάλιση, εξασφάλιση των παιδιών όπως έχουμε στη Γερμανία ανεξαρτήτως από το καθεστώς των γονιών τους. Εμείς ζητάμε συγκεκριμένα 500 ευρώ ανά παιδί ανεξαρτήτως μορφής οικογένειας και θα βγάζουν οι γονείς. Και μετά βεβαίω η αντιστάθμιση θα γίνει μέσω του φορολογικού συστήματος. Ο γονιός ο οποίος κερδίζει πάρα πολύ ε, θα πληρώσει ούτως ή άλλως μέσω των φόρων περισσότερα. Το σκεπτικό εδώ πέρα είναι να έχει οικογένεια ή με συγχωρείτε κοινωνία ευθύνη για την επόμενη γενιά και για τα παιδιά συγκεκριμένα. Για τους γονείς, για να πάμε προς την κατεύθυνση του Big Society, θα μπορούσαμε να έχουμε μια διαγενειακή συνεισφορά που θα μπορούσε να είναι παραδείγματο χάρη μέσω των κοινωνικών εισφορών, μια ιδέα. Το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι τι γίνεται με τις οργανώσεις φτώχειας. Εμείς είμαστε μέλος και έχουμε στενή επαφή με την Εθνική Διάσκεψη Φτώχειας και στο ευρωπαϊκό επίπεδο είμαστε μέλος και συμμετέχουμε και με... έχουμε κοινέ απαιτήσει όσον αφορά τη μείωση των φτώχειας. Προσπαθούμε επίσης να επηρεάσουμε τις ε, πολιτικές ε, απαιτήσει που τίθενται, π.χ. για το πώ η πολιτική τη φτώχεια θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερο βάρο στις γυναίκες ε, στα... και πλευρά δικαιωμάτων. Το τρίτο πλέγμα, το θέμα λεφτά ή υπηρεσίες, ε, όσον αφορά τα επιδόματα. για τις ελάχιστες δηλαδή παροχές αυτό είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και ανθρώπινης αξιοπρέπειας που μπορεί να ρυθμιστεί μέσω αυτών των κανονισμών. Δηλαδή, αν ένα συνταγματικό δικαστήριο, όπως έχει κάνει το γερμανικό και θεωρεί την εκπαίδευση ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, τότε δεν μπορεί να κάνει κάτι αντίθετο ένα κράτος. και μέσω ανταγωνισμού ή δεν ξέρω ποιο άλλο τρόπο να καταστήσει αδύνατη την παροχή μια τέτοια υπηρεσία. Δηλαδή, αυτό σημαίνει πω το κράτο είναι υποχρεωμένο για λόγου ανθρώπινη αξιοπρέπεια να διαθέσει αυτέ τι υπηρεσίε σε όλου. Και όσον αφορά τα παιδιά, αυτό σημαίνει, κατά την άποψή μα, πω και οι γονεί θα πρέπει να έχουν μια αυτονομία για να ξέρουν ποια μέτρα επιλέγουν για τα παιδιά τους και να μην έχουν μόνο περιορισμένες επιλογές από το κράτος. Αυτές δηλαδή που προωθούνται από το κράτος. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία με τις οργανώσεις φτώχειας. Πάρα πολλά κοινά σημεία έχουμε, αλλά για εμάς είναι σημαντική η προσέγγιση που βασίζεται στα δικαιώματα, να περιοριστεί δηλαδή η φτώχεια των παιδιών και των γυναικών. Varmt tack för de här svaren på frågeställningarna. Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως για τη συμμετοχή σας σε αυτή την ακρόαση και για την απάντησή σας στις διάφορες ερωτήσεις. Και τώρα σας δίνω το λόγο για να συμπληρώσετε. Ναι, κάποια από αυτά που υπόθηκαν για τις υπηρεσίες λόγου χάρη, εδώ δεν πρέπει να περιοριζόμαστε μόνο στις με μονομένε υπηρεσίε. Κάτι που είναι σημαντικό για τι μονογονεϊκέ οικογένειε είναι η στέγαση. Πολλοί ζουν σε κοινωνικέ, όπω λέγονται, κατοικίε, ενοικιαζόμενε κατοικίε προφανώ. Και αυτό βεβαίω επηρεάζεται ζωή των οικογενειών και ιδιαίτερα των παιδιών. Μια άλλη πολύ σημαντική υπηρεσία είναι η υποδοχή, η η συνοδεία, η παρακολούθηση των ε, μητέρων που αναζητούν εργασία. Διάβασα πρόσφατα στην εφημερίδα ότι στις Βρυξέλλες υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα που στοχεύει ακριβώς τις ε, νέες αυτές μητέρες, τις ανοιπαντρές που ψάχνουν δουλειά και θα έχουν πιο εύκολη πρόσβαση σε νηπιαγωγεία, σε σταθμούς για την φύλαξη των παιδιών Υπάρχουν ε, παραδείγματα όπως ε, αυτό του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την καταπολέμηση της φτώχειας που ασχολήθηκε πολύ με τα θέματα αυτά, ιδίως με την πρόσβαση στην ενέργεια. Η ενεργειακή φτώχεια είναι ένα στοιχείο που έχει τεράστιες συνέπειες για την ε, κατάσταση των μονογονεϊκών οικογενειών και ιδίως των παιδιών. Πολλά μπορούν να γίνουν ως προς την πρόσβαση στις υπηρεσίες. Για μας το ζήτημα δεν είναι κάτι φαίνεται αμεληταίο. Μπορεί να φαίνεται ελάχιστο όλο αυτό, αλλά το ελάχιστο εισόδημα που ανέφερε η κυρία Τόμψον είναι σημαντικό. Επιτέλους υπάρχουν στατιστικές, υπάρχουν αριθμητικοί στόχοι για την καταπολέμηση της φτώχειας μέχρι το 2020 όμως ακόμη μιλάμε για αριθμητικούς στόχους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη-μέλη όπως τους αρέσει. Γιατί υπάρχουν τρεις υποδείκτες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ε, να χρησιμοποιηθούν κατά τη βούληση του καθενός. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο λιγμών. Εν τέλει, Είναι σημαντικό να έχουμε στόχο με συγκεκριμένο ποσοστό μείωση της στόχης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά το θέμα είναι πώς αυτός ο, το ποσοστό, αυτό ο δείκτη θα υλοποιηθεί. Ευχαριστώ για αυτές τις συμπληρωματικές πληροφορίες. Αφήνω την Προεδρία και κυρίως το λόγο στην εισηγήτριά μας, στην κυρία Ματέρα, ώστε να ανακεφαλαιώσει την όλη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως σωστά είπατε, ως εισηγήτρια για την έκθεση αυτή, θα επικεντρωθώ κατά κύριο λόγο στην έγκαιρη και αποτελεσματική και συγκεκριμένη στήριξη των single mothers, των ε, ανήπαντρων μητέρων. Ακούσαμε τις συνεισφορές τόσων συναδέλφων που έθιξαν προβλήματα ή συσχετισμούς με άλλα προβλήματα, όπως η φτώχεια των παιδιών. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στις Επιτροπές του Κοινοβουλίου θα μπορέσουμε να επικεντρωθούμε στο συντακτικό τμήμα του όλου θέματος όπως πρέπει να κάνουμε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ όλες όσες παρενέβησαν, όλες τις εμπειρογνώμονες και όλες τις συναδέλφους. Διότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό να ε, μπορέσω να συγκρατήσω όλα αυτά που τόσο πυκνά σημείωνα, που με τόσο ενδιαφέρον άκουσα και να τα μελετήσω ήδη από τις επόμενες μέρες και ήδη η εργασία μας να ξεκινήσει κατευθείαν και να είναι και αποτελεσματική. Το να καταπολεμήσουμε την φτώχεια σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε τις δυναμικές που επικρατούν στο πλαίσιο των οικογενειών, της κοινωνικής πρόνοιας και της αγοράς εργασίας. Θα πρέπει να καταλάβουμε τις συνθήκες και την διακριτική μεταχείριση κατά των φύλων, όπως επηρεάζονται από τις οικογενειακές εξελίξεις και τις δημογραφικές εξελίξεις της κοινωνίας μας και τα εθνικά συστήματα. Ως τώρα έχουμε δει ε, πώ έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιστραφεί η πορεία. κάποιε φορέ δεν υπάρχει αρκετή κοινωνική πρόνοια, η προστασία είναι ανεπαρκής, δεν υπάρχει επαρκή κατάλληλο συνδυασμό επαγγελματικού και προσωπικού βίου. Ε, η, η μονογονεϊκή οικογένεια πολλέ φορέ σημαίνει ότι υπάρχει και ένα μόνο μισθό. Όλε αυτέ οι συνθήκε επιβαρύνουν και σημαίνει ότι μπορεί μια μονογονική οικογένεια να καταλήξει στην φτώχεια. Δεν σημαίνει επίση μια οικογένεια μονογονική ότι υπάρχει μια μαμά και ένα γιο, αλλά μπορεί να υπάρχουν περισσότερα παιδιά. Εδώ πρέπει λοιπόν να εμβαθύνουμε από την άποψη την κοινωνιολογική, την πρακτική, τη στατιστική και να δούμε τι συμβολέ μπορούμε να συγκεντρώσουμε από επιστήμονε, ερευνητέ που καθημερινά, μέρα με τη μέρα, από χρόνια συμβάλλουν στο έργο αυτό και μας δίνουν ε, μια κατάλληλη συνεισφορά όπου εμείς ως ευρωβουλευτές που εκπροσωπούμε το λαό 27 διαφορετικών χωρών στην συγκεκριμένη περίπτωση τα χρειαζόμαστε. Εγώ λοιπόν θα φροντίσω να τα λάβω υπόψη. Και για τις συγκεκριμένες λύσεις που προτάθηκαν μέσα από την εξέλιξη της συζήτησής μας ήταν σημαντικές. Ε, υποδομές για την φροντίδα των παιδιών με οικονομικές διευκολύνσεις και μορφές εργασίας πιο ευέλικτες, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα απασχόλησης και των παιδιών, να έχει κανείς και περισσότερα παιδιά μάλιστα και κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών να υπάρχει φροντίδα. Ε, επίσης οι νομικές ευθύνες των γονέων, των πατέρων, οι οποίοι μετά τον χωρισμό, το διαζύγιο δεν ασχολούνται πλέον όχι μόνο από οικονομικής άποψης, αλλά και από ηθικής πλευράς με τα παιδιά τους. Και έπειτα για τον χωρισμό των γονέων, το διαζύγιο. Πολλέ φορέ συμβαίνει, όπω το είπαν πολλέ φορέ οι συνάδελφοι και οι εμπειρογνώμονε, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, κάποιε φορέ υπάρχει επιδείνωση των συνδικών διαβίωση, άρα και κοινωνικό αποκλεισμό. Όχι μόνο των γυναικών, αλλά και των ίδιων των παιδιών. Έχουν δυσκολίε να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίε ε, ή η δυσκολία θα, θα μπορούσε να προκύψει στο κοινωνικό ιστό και θα πρέπει να του δοθεί δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά σε θέσει εργασία στην ίδια κοινωνία. Συνεχώ μιλάμε για βελτίωση, για εξακολούθηση ανάπτυξη και στα στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020 μιλάμε για τι μεγάλε ευκαιρίε που πρέπει να δώσουμε στου νέου. Ε, το συζητάει και η Επιτροπή Προπολογισμών. Το θέμα είναι πόσο επενδύουμε στη στρατηγική αυτή ε, και πόσο λαμβάνουμε υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία ενώ επικεντρωνόμαστε κατά τα άλλα στους νέους. Αυτά. Νομίζω ότι δυστυχώς δεν μπορέσαμε να συζητήσουμε σήμερα τα πολυάριθμα εμπόδια, τους φραγμούς που υπάρχουν και τα οποία εμείς ως εκπρόσωποι των πολιτών θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε αφού τα συναντούμε και Έχουμε και το πρόβλημα ότι η συνεισφορά μας δεν γίνεται πάντοτε αρκετά συγκεκριμένη και αποτελεσματική. Εμείς όμως ως εκπρόσωποι των γυναικών, των οποίων θέλουμε να προσπιστούμε τα δικαιώματα και την ισότητα των φίλων το ίδιο, θα πρέπει ως προς αυτό, ε, και εγώ και όλες οι συνάδελφοι που ξέρω ότι είναι ταγμένοι στον σκοπό αυτό όπως εγώ ίδια, θα πρέπει να είμαστε συγκεκριμένες ακριβείς να εντοπίζουμε αμέσως στόχο και να κοιτάζουμε πώς θα το πετύχουμε. Δεν θέλω να καθυστερήσω, θα σας δώσω εγώ ίδια τον λόγο από μόνη μου. Θα ήθελα να συνεχίσω τη συζήτηση αυτή, αλλά νομίζω ότι ο χρόνος ήδη ήταν με το πλευρό μας. Μιλήσαμε και συζητήσαμε αρκετά. Δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε. Τη δουλειά θα την ξεκινήσω ήδη από σήμερα και σας ευχαριστώ που ήρθατε και είχατε τόσο μεγάλη προσέλευση. Νομίζω λοιπόν ότι ολοκληρώσαμε κιόλας, έτσι. Ωραία λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Ματέρα και κυρία Ματέρα στα συμπερασματά της μίλησε για την οικονομία, τις επενδύσεις και στην Επιτροπή Προπολογισμού και τα λοιπά. Και άρα μπορώ και εγώ να πω πως πιο σημαντική επενδύσεις θα κάνουμε στο μέλλον είναι η επένδυση στα παιδιά. Νομίζω το να ξέρουμε την αξία των παιδιών και την αξιοπρέπεια των παιδιών και το ότι όλα τα παιδιά έχουν ίσα δικαιώματα, το δικαίωμα να μεγαλώσουν σε μια κοινωνία όπου ε, γίνεται σεβαστή αξιοπρέπεια όλων των παιδιών, όλα τα παιδιά έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, να μεγαλώσουν, να απτυχθούν στην κοινωνία. Αυτή είναι η καλύτερη δυνατή επένδυση που μπορούμε να κάνουμε. Είναι πολύ καλό το να τελειώνουμε τη σημερινή συζήτηση με αυτό το πνεύμα. Ε, ότι δηλαδή οι ευκαιρίες δηλαδή των παιδιών είναι βασικό κομμάτι της πολιτικής μας και βεβαίως αναμένουμε τη συνεργασία μας με την κυρία Ματέρα στο μέλλον και τις κοιοδησηγήτριες έτσι ώστε η γνωμοδότηση να είναι όσο δυνατόν καλύτερη μπορεί να είναι. Είναι λοιπόν σημαντικό το θέμα, θα συνεχίσουμε την εργασία μας. Χαίρομαι που είχαμε αυτή την ευκαιρία σήμερα να ακούσουμε και το οποίο είχαν να μας πούν οι προσκεκλημένες μας και σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα και ευχαριστώ και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνεισέφερε. Ευχαριστώ την κυρία Ματέρα, ευχαριστώ τις συναδέλφους, ευχαριστώ τη γραμματεία. για το ότι κατέστησαν δυνατή τη σημερινή ακρόαση. Ευχαριστώ και τους Ερμηνείς που μας επέτρεψαν να συνεννοηθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.